Ladies and gentlemen, good morning. Please be seated. Παρακαλώ, καθίστε, συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο θέμα και την κυρία Βαλέρο εδώ. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε με το εργαστήριο ήθελα να ξεκινήσουν οι πράσινοι και η κυρία Βαλέρο η ίδια θέμα είναι η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου εξαγωγών όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαρά καλωσορίζω την κυρία Σίδλα Μπάουερ, την δόκτορα Σίδλα Μπάουερ, ε, ερευνήτρια του γνωστού και μη εξαιρετέου Ινστιτούτου της Στοκχόλμης ε, του Κύπρη. Το θέμα είναι γνωστό. Το έχουμε συζητήσει ήδη σε πολλές ε, συνεδριάσεις. Ε, είχαμε και ενημέρωση. Οπότε θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Μπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που με κάλεσε να μιλήσω και να συνεισφέρω και εγώ στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους έλεγχους εξαγωγών και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εδώ και πολλές δεκαετίες από δεκαετία του 90 παίζει πολύ ενεργό ρόλο. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό στο οποίο ε, έκανα την πρώτη μου σχετική εκδήλωση πριν από 20 χρόνια. 20 χρόνια το Νοέμβριο του 97. Και έκτοτε παρακολουθώ το ζήτημα αυτό και οφείλω να πω ότι δεν το βαριέμαι ποτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει δραστήριο. Πριν ξεκινήσω να πω δύο πράγματα για το ΣΥΠΡΙ. Νομίζω πως περισσότεροι θα ξέρετε το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης. Να σας πω ότι ιδρυθήκαμε το 1966 ακριβώ για να τιμήσουμε τα 150 χρόνια της ε, διάληπτης ειρήνης ε, στην Σουηδία. Είμαστε υπερκομματικό Ινστιτούτο, το οποίο ίδρυσε το Κοινοβούλιο της ε, χώρας και στόχο έχουμε ακριβώς να προωθούμε την συζήτηση του αφοπλισμού. Η ιδέα ανήκε στον κύριο Μύρνταλ, ο οποίος ήταν πρέσβης τότε στην Γενέβη της Σουηδίας και βεβαίως ε, είχε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοια στοιχεία. Όλοι βεβαίως ε, γνωρίζετε τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή θέση, το έγγραφο το οποίο υπάρχει από το 2008. Αλλά για να υπενθυμίσω Υπάρχουν ε, πέντε κύρια στοιχεία, τα οχτώ κριτήρια μαζί με τον οδηγό χρήστη που αφορούν την εφαρμογή. Υπάρχουν μηχανισμοί για ανταλλαγή πληροφοριών, μηχανισμοί επιβολής, ε, αναφοράς ε, και όλα αυτά σχετίζονται με έναν κοινό κατάλογο υλικού πολέμου. Τώρα αυτά τα έχουμε συνηθίσει βεβαίως, αλλά 20 χρόνια πριν δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Ήταν καινοτόμα επαναστατικά τολμώ να Και επίσης παρά το ότι σε γενικές γραμμές μιλάμε για τις εξαγωγές όπλων, ε, η κοινή θέση είναι ευρύτερη γιατί αφορά και την μεταφόρτωση και την ε, διαμεσολάβηση και τη μεταφορά τεχνολογίας ε, και software και παραγωγής κατόπιν αδείας. Οπότε είναι ευρύτατο μέσο. Επίσης, για να δούμε τη σημασία αυτού του μέσου, όταν δούμε τα νούμερα του Διεθνούς Εμπορίου Όπλων είναι πολύ σημαντικά και αν δείτε τα στοιχεία του ΣΥΠΡΙ για το διεθνές ε, εμπόριο όπλων, συμβατικών όπλων, οι πέντε μεγαλύτεροι εξαγωγείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 20% των εξαγωγιών τα τελευταία πέντε χρόνια. Οπότε η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ρύθμιση και τον έλεγχο αυτών των αγαθών είναι ε, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και για να επαναλάβω ποιοι είναι οι πέντε μεγαλύτεροι εξαγωγείς ε, της Ένωσης. Είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία. Και κάποιες άλλες χώρες βεβαίως παράγουν όπλα και τα εξάγουν. Οπότε, για να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου εξαγωγής όπλων. Θα ξεκινήσω με μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ε, και μετά θα δώσουμε κάποιες επιλογές για το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Λογικά λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια κοινή θέση, Έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Και μάλιστα αν το βέλγικο σύστημα, ε, έχουμε 30 τέτοια συστήματα. Δηλαδή τα διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες παίζουν διαφορετικό ρόλο. Αλλού μπορεί να είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλού το Υπουργείο Οικονομίας ή μια ανεξάρτητη αρχή αλλού έχουν βέτο τα Υπουργεία, αλλού έχουν ένα συμβουλευτικό ρόλο. Όλα θα λοιπόν εξαρτώνται από χώρα σε χώρα. Επίσης υπάρχουν πολύ σοβαρές διαφορές όσον αφορά την δυνατότητα αναστολής ή αφαίρεσης αδείας. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην Αυγική Άνοιξη όταν ε, πολλές ε, χώρες ε, μετάνιωσαν για την άδεια εξαγωγών και προσπάθησαν να ανακαλέσουν άδειε για εξαγωγέ που δεν είχαν φύγει από τη χώρα. Και βέβαια υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία των κριτηρίων, κάτι το οποίο αναφέρεται συχνά είναι το κριτήριο 8, το οποίο αφορά την ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην συνθήκη αυτή, στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε μια άτυπη συνάντηση των ε, μερών στη Γενέβη την Παρασκευή και ο πρόεδρος ε, που είναι Φιλανδός έθεσε το ζήτημα μεταξύ της συνθήκης αυτής ε, και των αναπτυξιακών στόχων στην ημερήσια διάταξη. Οπότε το συζήτησαν ένα ολόκληρο απόγευμα για τη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το κριτήριο αυτό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μετά έχουμε τον οδηγό χρήστη που πολλοί θα έχετε μελετήσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο παρελθόν υπήρχαν μόνο τα κριτήρια βοήθειας, τα, τα 8 κριτήρια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Οπότε με τον οδηγό των Χριστών υπήρχε μια συνένεση για τον τρόπο ερμηνείας και για το ποιε πηγές ε, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των κριτηρίων. Επίση, έχουμε πολλές πληροφορίες ε, στο πλαίσιο της κοινή θέση μεταξύ κρατών μελών για άδειε που έχουν απορριφθεί, κάτι το οποίο υπήρχε εξ αρχής, αλλά όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουν εκδοθεί, είναι πολύ πιο λίγες οι ανταλλαγές πληροφοριών. Οι πληροφορίες μοιράζονται. Είναι στο πλαίσιο ενός tour de table ε, σε σχέση με κάποιες χώρες ε, που λαμβάνουν την βοήθεια, αλλά κατά τα λοιπά ε, οι πληροφορίες υπάρχουν στην ετήσια έκθεση που ξέρετε πως πάντα είναι εκ Αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι μια βελτίωση στο πληροφοριακό σύστημα για να μοιράζονται πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Ήταν ένας ε, μηχανισμός, ε, ένα CD που μοίραζαν με πληροφορίες, τα σαν έχουμε προχωρήσει έκτοτε. Ε, και έχουμε ένα σύστημα πληροφοριακό για να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Λοιπόν, κάποιες από τις επιλογές ε, τώρα ενίσχυσης και εφαρμογής της κοινή θέση. Μία δυνατότητα είναι να κάνουμε κάτι το οποίο έχει γίνει νομίζω επιτυχώς όσον αφορά τον κανονισμό που είναι μία διαδικασία αξιολόγησης ε, από μοτίμους όπου μπορούν τα κράτη-μέλη να ανταλλάξουν επισκέψεις στις πρωτεύουσες και να κοιτάξουν κάποιες πτυχές ε, και να δουν πώς εφαρμόζονται λεπτομερώς ε, οι διατάξεις αυτές. Οπότε οι αρμόδιοι για το θέμα και οι και αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τα σχετικά. Και βεβαίως καλό είναι να δουν και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των 8 κριτηρίων, γιατί αυτό το είχαμε μελετήσει πριν από λίγα χρόνια και ρωτήσαμε εξ ονόματος μιας χώρας πώς ακριβώς εφαρμόζονται τα κριτήρια, δηλαδή αν θέλουν να ε, αξιολογήσουν την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα, ποιες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν, ποιες ερωτήσεις γίνονται στον αρμόδιο στο Υπουργείο Εξωτερικών και οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ε, πρώτον πολύ διαφορετικές και δεύτερον καταλάβουμε ότι μια χώρα δεν είχε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή κάποιες αξιολογήσεις ήταν λίγες λέξεις, άλλες ήταν ολόκληρο μυθιστόρημα. Οπότε και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης ανέφερα ότι γίνεται ένας γύρος τραπέζης ε, στις ε, συναντήσεις για κάποιες χώρες οι οποίες λαμβάνουν βοήθεια και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο μέσο που ίσως ε, θυμάστε αφορά ακριβώς την εργαλειοθήκη για μετά τα εμπάρκο που είχε συζητηθεί το 2004 μετά την άρση του εμπάρκο της Λιβύης τότε και ήταν ένα πολύ εξαιρετικό μέσο ε, δυστυχώς ε, έμπλεξε με την συζήτηση για το εμπάργο κατά της Κίνας και δεν υιοθετήθηκε ποτέ επισήμως. Οπότε Καλό θα ήταν να επανέλθει αυτό γιατί προέβλεπε μια τρίμηνη ανταλλαγή πληροφοριών για τέτοια ζητήματα που αφορούσαν παραδείγματο χάρη τον τύπο εξοπλισμού, τον τελικό χρήστη και επίσης τακτικές διαβουλεύσεις και συζητήσει στο επίπεδο του Συμβουλίου αν υπήρχε κάποια αλλαγή πολιτικής. Οπότε αν είχαμε ένα τέτοιο μέσο είτε για χώρες ε, μετά από ένα εμπάργκο, είτε για ευαίσθητες φορές για τις οποίες δεν συμφωνούν όλα τα κρατημέλη. Νομίζω πως αυτό θα ήταν κάτι το σημαντικό. Επίσης υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσαν να μοιραστούν τα κρατημέλη. Π.χ. σε περίπτωση όπου καταλήγουν αλλού τα όπλα σε πλαστά πιστοποιητικά, σε ύποπτους διαμεσολαβητές ή εταιρείε μεταφορών και σε άδειες που έχουν ανασταλεί ή ε, αποσυρθεί. Και δύο άλλες επιλογές που θέλουμε να δούμε είναι για να ενισχυθεί η κοινή θέση και αυτό μάλλον ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο που είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι μπορεί να ενισχυθεί η διατύπωση της κοινή θέση γιατί αυτή τη στιγμή μια, μια αξιολόγηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά πάντα υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ αυτών που βλέπουν μια λειτουργική, μια προσέγγιση λειτουργική και αυτών που θέλουν μια προσέγγιση αρχών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή η χρήση του συγκεκριμένου όπλου σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αξιολογούμε γενικότερα την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα και τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές θέσεις. Και βεβαίως έχουμε και τον οδηγό ε, χρήστη που είναι πάρα πολύ χρήσιμος αλλά είναι ένα έγγραφο PDF και στον σημερινό κόσμο μπορεί να γίνει πολύ πιο φιλικό προς τον χρήστη και να γίνει ένα πιο διαδραστικό εργαλείο. Πάμε τώρα στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Στην κοινή θέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να ενισχύσει την παροχή πληροφοριών για τις εξαγωγές όπλων. Και να υπενθυμίσω σε όλους όσους έχουν δει την πρώτη πρώτη έκθεση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Διοντολογίας που ήταν μονοσέλιδος. Ε, ήταν μεγάλο επίτευγμα και τότε χρειάστηκε μεγάλη πίεση από τη Φιλανδική Προεδρία ούτως ώστε να δημοσιευθεί αυτή η μία σελίδα. Σήμερα έχουμε εκατοντάδες σελίδες ε, εκατοντάδες σελίδων εκθέσεις, δηλαδή έχουμε αλλάξει πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά περιφορία βελτίωσης. Εδώ στη γραφική παράσταση βλέπετε ότι δεν έχουμε όλα τα κράτη-μέλη που, κάνουν, που υποβάλλουν πλήρες εκθέσεις. Πλήρες εκθέσεις σημαίνει ότι έχετε, δίνετε πλήρες πληροφορίες και για τις ε, άδειες που εκδίδετε, αλλά και για τις πραγματικές παραδόσεις όπλων τα πραγματικά νούμερα. Και υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι γι' αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να τους ψάξουμε. Μερικές φορές ε, δεν υπάρχουν, υπάρχουν αρκετά θέματα, αρκετά προσωπικό, μερικές φορές ε, υπάρχει θέμα μυστικότητας, μερικές φορές ε, υπάρχουν θέματα προτεραιότητας πολιτικής. Ε, δεν υπάρχει κατάλληλη πληροφορική πολλές φορές για να δώσετε τις πληροφορίες. Και πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα αυτό που μπορεί να επιληθεί. Ε, Τώρα, συνοψίζω την κατάσταση για τις υποχρεώσεις υποβολή εκθέσεων. Όταν βλέπετε τον αριθμό των κρατών μελών που, κάνουν πλήρες, που υποβάλλουν πλήρε εκθέσεις, φτάσαμε ε, από τα 28 κράτη-μέλη σε ένα μέγιστο νούμερο 21. Μετά πέσαμε στα 20. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι για τα μεγάλα κράτη όπω η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι δεν μπορούν να δώσουν λεπτομερεί πληροφορίε για τι πραγματικέ εξαγωγέ όπλων. Οι χώρε, όπω η Σουηδία αλλά και άλλες που δίνουν τέτοια λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία τα παίρνουν κυρίως από την ε, βιομηχανία, τον κλάδο που είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ε, νούμερα για το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν τις άδειε που έχουν λάβει. Και επίσης ε, παίρνουν ε, αυτά τα νούμερα και από τελωνιακά, τελωνιακές πηγές. Πολλά κράτη-μέλη όμω δυσκολεύονται πάρα πολύ σε αυτό. Και πιστεύω ότι παρότι φαίνεται το πρόβλημα να είναι τεχνικό, ε, Νομίζω ότι αν θεωρηθεί πολιτική προτεραιότητα θα μπορούσε να λυθεί ακόμα και με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων και με τη βοήθεια εδώ των Βρυξελών που θα μπορούσε να βοηθήσει για να δώσει ε, τις, τους κατάλληλους σχετισμούς, ε, τύπους κτλ. για τα όπλα. Ε, μερικές φορές υπάρχει το επιχείρημα ότι οι άδειες είναι το πραγματικό, η πραγματική πληροφορία. Γιατί χρειαζόμαστε και πραγματικές, ε, πραγματικά νούμερα για τις πραγματικές εξαγωγές όπλων. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά έχουμε ανοιχτές άδειε, όπου πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο πραγματικός όγκος ε, των εξαγωγών, ε, ούτε καν τον ε, και των εγκρίσεων που έχουν δοθεί. Και τελικά πόσα όπλα φτάνουν στην ε, χώρα παραλαβής. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ο χρονισμός Οπότε υποβάλλεται η έκθεση συχνά, ε, υποβάλλεται αρκετά αργά. Ένα χρόνο μετά από την στιγμή που παραδόθηκε η τελευταία παρτίδα όπλων. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο, μεγάλο κενό ανάμεσα ε, στη χρονική στιγμή που ελήφθη η απόφαση μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει το Κοινοβούλιο να ελέγξει τα στοιχεία. Προχωράμε στις επιλογές που έχουμε για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Καταρχάς, Υπάρχουν διάφορα βήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν και να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να υποβάλουν πλήρε εκθέσει ε, για την ετήσια δικές εκθέσεις για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε να, καταρχάς μπορούμε να εμπνευστούμε από τις χώρες που δίνουν πραγματικά νούμερα ε, και να εμπνευστούν κυρίως οι χώρες που λένε ότι τεχνικά δεν είναι δυνατόν αυτό. Ε, και θα μπορούσε να γίνει και συζήτηση σε υψηλότερο επίπεδο ε, να συνεργαστούμε ας πούμε, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων, δημιουργώντα κώδικε που θα μα επέτρεπαν να ανοιχνεύσουμε και να αναζητήσουμε τι πληροφορίε από τι βάσει δεδομένων τελωνίων. Και για να είναι πιο επίκαιρε αυτέ οι εκθέσει, πολλά μπορούν να γίνουν. Καταρχά, ένα προφανέ είναι να έχουμε μια ε, άλλη προθεσμία, ε, πιο σφιχτή για την υποβολή των εκθέσεων των κρατών μελών, αλλά ακολουθώντα και αυτά που έκαναν κάποια κράτη-μέλη, να έχουμε περισσότερε από μία αιτήσει εκθέσει. Ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν μηνιαίε, όπω η Ολλανδία, μηνιαίε εκθέσει. Ε, και άλλοι, όπω η Γερμανία, ε, έβαλε πρόσφατα την υποχρέωση υποβολή ε, εξαμηνιαίων εκθέσεων. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πολλά για να υποβάλουν οι εκθέσει πιο εγκαίρω και να είναι πιο επίκαιρε. Τι πέτυχε ακόμα η θέση τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για πρώτη φορά ε, υπάρχει ένας κανόνας για την, ε, τις εθνικές εκθέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα κρατημέλη ενθαρρύνονται να ετοιμάζουν ε, μια εθνική έκθεση για τις εξαγωγές όπλων και από τη γραφική παραστασία που βλέπετε φαίνεται ότι το ποσοστό ανέβηκε πάρα πολύ. Αλλά μόνο τα τρία τέταρτα των κρατών μελών δημοσιεύουν αυτή την ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων. Και ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό να έχουμε μια συμπληρωματική έκθεση, εθνική έκθεση δηλαδή για τις εξαγωγές όπλων πέρα από την ε, ενωσιακή, είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις λογοδοτούν στα εθνικά τους κοινοβούλια, που χρειάζονται λεπτομέρειες πληροφορίες για να αξιολογήσουν ε, το πώς ε, ελήφθησαν οι πολιτικές αποφάσεις. Και ένας από τους λόγους που αυτό είναι σημαντικό είναι ότι φυσικά, η, λογικά, οι εξαγωγές όπλων ε, είναι αντικείμενο ε, συγκρουόμενων ε, συμφερόντων. Υπάρχουν θέματα αμυντικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, ακόμα υπάρχουν και επιχειρήματα αντικατασκοπίας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Καταπολέμηση λοιπόν της τρομοκρατίας που έχουμε φτάσει, υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη των συγκρούσεων, και τα θέματα της ανάπτυξης. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα, όλα αυτά τα συμφέροντα δεν πηγαίνουν προς την ίδια Θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να σταθμίσει τους παράγοντες αυτούς και να κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου που να βασίζεται και στην πρόβλεψη για το μέλλον. Κανένα δεν ξέρει απόλυτα για το πώς ε, θα εξελιχθεί η κατάσταση στη χώρα που εισάγει τα όπλα. Επομένως, το αποτέλεσμα της ε, αξιολόγησης αυτής είναι ότι όλες αυτές οι παράμετροι απεικονίζονται στην εθνική έκθεση. Μερικές φορές υπάρχουν τα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας που οδηγούν στο να παραδοθούν περισσότερα όπλα παρά να περιοριστούν. Αλλά εμείς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Και ένας από τους λόγους που υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1992 τα κριτήρια βοήθειας είναι ε, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι άμα παραδοθούν αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τελικά εναντίον των δικών σου ε, ενόπλων δυνάμεων. Ε, Επομένω, για λόγου ασφάλεια, κάποιε εξαγωγέ όπλων καλό είναι να μην γίνονται. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε όχι μόνο τα θέματα του χρονοδιαγράμματος ε, για την υποβολή εκθέσεων, αλλά και το κενό που σας ανέφερα, το χρονικό κενό, αλλά και τις ε, διαθέσιμες πληροφορίες μετά. Και βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιο χρονικό διάστημα ε, από τη στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις μέχρι να ε, δημοσιευθούν οι πληροφορίες και να συζητηθούν από το κοινό και από τα κοινοβούλια. Και τώρα προχωράμε στις δυνατότητες που έχουμε για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα, ορισμένα τα ανέφερα ήδη και δεν θα τα σχολιάσω λεπτομερώς, αλλά θέλω να πω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πολλές από τις πληροφορίες που δίδονται ακόμα και σε μια πολύ πολυσέλιδη έκθεση δεν σου επιτρέπουν να αξιολογήσεις το πώς έχουν εφαρμοστεί τα κριτήρια. Και νομίζω ότι το ξεχνάμε αυτό το σημαντικό σημείο, ότι συχνά οι κυβερνήσεις βάζουν τις πληροφορίες μέσα στην έκθεση που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη οι πληροφορίες που χρειάζεσαι ως ε, πολίτης ή ως ε, βουλευτής στο Κοινοβουλίο για να απαντήσεις σε ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εγώ αυτό που θα πρότεινα λοιπόν είναι να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή να λέμε να ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί και να ποιε είναι οι πληροφορίε που χρειάζομαι για να απαντήσω στην ερώτηση. Φερρυπίν, συχνά υπάρχει εστίαση σε αυτές τις εκθέσεις στην ε, αξία των αδειών, στην τιμή των αδειών. Καλές είναι οι στατιστικές, γιατί είναι εντυπωσιακέ για τις εφημερίδες και οι εφημερίδες αναφέρονται σε αυτό, αλλά ο πραγματικός, ε, η πραγματική αξία των εξαγωγών στις τρίτες ε, χώρες, αν λάβεις υπόψη σου μόνο αυτό το στοιχείο, τα χρήματα δηλαδή, αυτό, από αυτό δεν βλέπεις ε, το πόσο έχουν βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό έχει σημασία και από το ποιος είναι ο τελικός χρήστης, ε, το είδος των όπλων, τον πραγματικό όγκο των όπλων κτλ. Συχνά όμως τα τελευταία χρόνια εστιάσαμε μόνο στο θέμα του όγκου ας πούμε, των όπλων, α, του αριθμού των όπλων, αλλά όχι στα υπόλοιπα βασικά σημεία. Ένα από τα πράγματα που θα μπορούσε να αλλάξει για να γίνουν οι, ευρω... εκθέσεις πιο διαφανείς ε, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν να δούμε τι είδη όπλων έχουν παραδοθεί σε, ποιον και πώς ε, επηρεάζονται τα κριτήρια που αφορούν την ε, βοήθεια. Επίσης, ποιο είναι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στα 28 κράτη-μέλη. Όταν δει το ρόλο και το συγκρίνει. Βλέπει ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Ορισμένα κοινοβουλία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τι εξαγωγέ όπλων, ορισμένα καθόλου. Μερικά, όπως ε, η Σουηδία, έχουν και μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που λαμβάνει και πληροφορίες για τις εξαγωγές όπλων πριν ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Και αλλού, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, λαμβάνεται από το Κοινοβούλιο η απόφαση, η ενημέρωση ε, η ενημέρωση μόνο αφού ληφθεί πολιτική απόφαση, αλλά ε, ελέγχουν πάρα πολύ ε, το θέμα της αδειοδότησης. Και στη Γερμανία και στην Ολλανδία πρόσφατα έλαβαν βήμα αποφάσεις για να, δώσουν, να δίνουν πληροφορίες πολύ πιο νωρίς στο Κοινοβούλιο. Τώρα το Κοινοβούλιο λοιπόν στις δύο αυτές χώρες λαμβάνει τις πληροφορίες λίγες εβδομάδες μετά, ενώ παλιά τις λάμβανε μήνες μετά ή και χρόνια μετά. Επομένως, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά για να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών, αλλά και ο ρόλος των κοινοβουλίων στον έλεγχο. Άρα, τώρα να δούμε τι έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, ούτως ώστε να βελτιωθεί το κείμενο να αλλάχτούν, να, ποιε πληροφορίε είναι, να μεταβληθεί αυτό, να συμπληρωθούν οι πληροφορίες και να γίνεται πιο ενδελεχής περιγραφή, ποια είναι τα προϊόντα, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ε, τι γίνεται όσον αφορά το, το στρατό και άρα να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες γενικότερα οπότε να προσεχθεί επίσης το θέμα των πιο σημαντικών συναλλαγών και όχι πιο επίμαχες ε, ε, πιο επίμαχοι προβληματισμοί. Επίσης θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις ούτως ώστε να είναι πιο εύχριστο το κείμενο ας πούμε να υπάρχουν έγγραφα σε PDF να υπάρχουν κάποιο είδους βάσεις δεδομένων που να είναι interactive και άρα θα μπορούσαμε πολλά να κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση επίσης διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας αλλά έχουμε και σημαντικές εξαγωγές, αλλά η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εποπτεία των εξαγωγών είναι πολύ περιορισμένη. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινοβουλίων. Και τώρα τελευταία αλλά σημαντικά κάποια θέματα όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Βελτιώσει θα μπορούσε να υπάρξει στους ε, ελέγχους και στην επιμελητία. Δηλαδή, τα μικρότερα κράτη-μέλη δεν έχουν παντού πρεσβείες. Άρα για τα μικρότερα κράτη-μέλη τον έρθουν σε επαφή είναι πιο δύσκολο ας πούμε για να ελεγχθεί μια διεύθυνση αν υπάρχει η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ή άσκηση κάποιου ελέγχου σε κάποια παράδοση όπλων. Τα μεγαλύτερα κρατημέλη μπορούν να τα κάνουν αυτά, αλλά μιλούμε για ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, στη Γερμανία, τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Ε, πολλές φορές είναι και θέμα εθνικής κυριαρχίας, αλλά θα πρέπει κανείς να συμφωνήσει για μια σύμβαση με την χώρα ε, όπου προορίζεται ένα φορτίο όπλων. Οπότε τώρα θα μπορούσε να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια χρειάζεται σχετική εκπαίδευση. Γιατί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και διπλωμάτες, αλλά με διπλό τρόπο πρώτα-πρώτα. Υπάρχει το θέμα του ελέγχου και του αν κάποιος έχει το τεχνικό background και από την άλλη μεριά για το θέμα κάποιες παράδοσες θα πρέπει τελικά κάποιος να ξέρει πέντε πράγματα. Οπότε θα, θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να κινηθούμε αλλά και κάτι άλλο που θα πρέπει να δούμε είναι αυτή η κατάτμιση του καθεστώτος ελέγχου. Αυτό ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τι γίνεται όσον αφορά τις εξαγωγές, αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλου είδους νομοθετήματα κοινοτικού δικαίου, τα οποία σχετίζονται με το θέμα. Ο κανονισμός για τα προϊόντα διπλής χρήσης, αυτό έχει να κάνει και με τα κριτήρια, την κοινή θέση επίσης. Την διαμετακόμιση των όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εμπάρκο των όπλων, ο καονισμός για τα πυροβόλα όπλα και είναι θέμα επίσης και αρμοδιοτήτων θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα μπορούσαν να εκτελεθούν προσπάθειες και για συντονισμό και για περισσότερη συνοχή, συνεκτικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μπορεί να το ενθαρρύνει και έτσι να δούμε πώς ο έλεγχος στις μέρους πολιτείας μπορεί να ε, γνωρίσει περισσότερο συντονισμό και επίσης να υπάρξει συνδυασμός των ε, επιμέρους προβληματισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα όπλα. Εδώ θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, αλλά να σας τονίσω τώρα καταληκτικά κάτι συγκεκριμένο. Το θέμα των πόρων. Γιατί και εδώ το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο. Από τη μια μεριά έχουμε το πόσοι ασχολούνται με τις εξαγωγές των όπλων. Το προσωπικό επ' αυτού είναι πολύ περιορισμένο. Είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένη η σύνθεση των ομάδων που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ε, επίσης, και ε, κάποιος προϋπολογισμός που αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων για τον έλεγχο των όπλων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι θετική εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν να προσφέρουν σημαντικά. Άρα θα πρέπει και εδώ να εκταμιευτούν πόροι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τελικά αυτή την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών. Σας ευχαριστούμε, δόκτωρα, για την παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω τον λόγο συναδέλφους και ε, πρώτα απ' όλα βεβαίως η κυρία Βαλέρο έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας παρουσίαση και για τις ιδέες που θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε στη νέα μας γνωμοδότηση το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω είναι ε, αν έχουν υπάρξει αλλαγές από την Αραβική Άνοιξη στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη πουλάνε όπλα και δίνουν άδειε στις χώρες εκείνες που είναι προβληματικές όπως η Σαουδική Αραβία χώρες ε, οι οποίες εμπλέκονται σε πραγματικό πόλεμο στην Ιεμένη. Έχουν υπάρξει έκτοτε αλλαγές. Να ε, μιλάω για τις νέες άδειες εξαγωγών. Και επίσης υπάρχει το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν ε, στοιχεία για το ποιες χώρες ακριβώς χρησιμοποιούν αυτό το κριτήριο για να απορρίψουν άδειε. Νομίζω πως υπάρχουν ελάχιστες χώρες ε, που χρησιμοποιούν αυτό το κριτήριο. Τώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλον για το πώς γίνεται η υποβολή εκθέσεων. Και την ε, τελευταία φορά βεβαίως ε, ε, είχε γίνει αυτό στην Επιτροπή αλλά εξαφανίστηκε στην Ολομέλεια. Πώς μπορούμε να κάνουμε το ζήτημα αυτό λιγότερο ευαίσθητο έτσι ώστε όλοι να πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις. Είναι όμως πολύ ευαίσθητο. Και στην τελευταία έκθεση εγώ ζήτησα εγώ έλαβα ε, επιστολή από την κυβέρνησή μου που μου έλεγε ε, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Χοντρικά, έτσι αυτό έλεγε. Ε, κάποιες χώρες απλά δεν υποβάλλουν εκθέσεις. Είναι λοιπόν και αυτό σημαντικό θέμα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής ε, κριτηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά ακριβώς το ερώτημα είναι εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά για την ε, καταπίεση του ίδιου του πληθυσμού της χώρας. Κάποιες χώρες κοιτάνε τη συνολική κατάσταση μιας χώρας, ενώ άλλες όχι. Ποιες χώρες κοιτάνε τη συνολική κατάσταση. Νομίζω ότι η Σουηδία το κάνει. Mm. Το γράφει νομοθεσία μας Βέβαια οι Σουηδοί έχουν μειώσει το επίπεδο απαιτήσεων. Θέλω να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τις άλλες χώρες. Πόσες ε, χώρες ε, έχουν σκεφτεί τη συνολική κατάσταση στην χώρα. Ήδη μας δώσατε πάντως πολλές ε, πληροφορίες, πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκάλερ, ε, θέλετε τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή έποψη της ε, κατάστασης. Βέβαιως, υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές προφανώς και αν δει κανείς ε, και συγκρίνει τις διάφορες καταστάσεις νομίζω πως εντάξει όταν υπάρχει εμπάργκο του ΟΗΕ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά μιας χώρας ε, υποθέτουμε ότι ακολουθείται μια κοινή ε, πρακτική. Εντάξει, αυτά είναι επίσημες αποφάσεις. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν χώρες οι οποίες από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριφέρονται λάθος και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ε, όπου ασκούμε κριτική στο α ή στο β. Ε, βλέπετε ας πούμε συμπεριφορά όπου παρά το ότι ασκούμε κριτική σε κάποιες χώρες παρόλα αυτά γίνονται εξαγωγές και ε, τα συζητάμε ε, και καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Π.χ. απέναντι στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχουν επίσημες αποφάσεις για εμπάργο όπλων. Είναι σαφές, αλλά κάποιες πολιτικές ε, της Σαουδικής Αραβίας νομίζω έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής και υπάρχει διαφορετική πρακτική. Ε, υπάρχουν κάποιες αιτιολογήσεις ε, το ερώτημα είναι μετά βεβαίως πώς ε, αντιδρούμε έτσι, από κοινού και το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι μήπως θα ήταν αποτελεσματικότερο να υπήρχε μια κοινή ε, αντίδραση Ναι, ίσως ε, και μέσω των ε, εθνικών ε, κοινοβουλίων. Αν μια συγκεκριμένη χώρα στέλνει τους πρέσβεις της στα εθνικά κοινοβούλια γιατί βεβαίως οι εθνικές κυβερνήσεις εμάς εδώ μας θεωρούν αδιάφορους ή ασήμαντους αλλά αν ε, είχαν παρόμοιες πρωτοβουλίες ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια, νομίζω πως αυτό θα ήταν πιο αποτελεσματικό σε μια πιο περιοριστική πολιτική. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν είμαι γενικά κατά των εξαγωγών όπλων. Και αν πραγματικά υπηρετεί τα πολιτικά μας συμφέροντα, είμαι υπέρ. Αλλά έχουμε και εκ των υστέρων, που βεβαίως είναι πάντα πολύ πιο εύκολο, ε, εμπειρίες ε, που βρεθήκαμε στη λάθος πλευρά. Ε, θα πρέπει νομίζω να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από κοινού για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ο τρίτος συντονιστής είναι ο κύριος Φανόρντεν. Θέλετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. και νομίζω όλοι συμφωνούμε στην ε, αδειοδότηση επικίνδυνων εμπορευμάτων, είτε μιλάμε για φάρμακα, είτε για όπλα. Αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο των ελέγχων εξαγωγών όπλων είμαστε πάρα πολύ καλοί στην ήπια νομοθεσία, την ήπια κριτική και τον ήπιο έλεγχο. Το ερώτημά μου είναι ε, το εξή. Ε, μήπως η απαγόρευση εξαγωγής, ε, ε, σε ποιες περιπτώσεις μάλλον η απαγόρευση εξαγωγής δυτικών όπλων είχαν θετικό αποτέλεσμα σε κάποια σύγκρουση στον κόσμο. Γιατί βλέπω πως υπάρχει ένας κλάδος ελέγχου εξαγωγών όπλων. Με μεγάλη περηφάνεια μιλήσατε για το ότι η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί από μία σελίδα σε εκατοντάδες σελίδες, σαν αυτό από μόνο του να αποτελούσε κάποιο επίτευγμα. Τι αποτέλεσμα όμως έχουν όλα αυτά στην πράξη, πέρα από το ότι κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα. Η Ρωσία και η Κίνα είναι δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων του κόσμου. Εξάγουν όπλα στους κακούς τι έλεγχοι υπάρχουν για αυτές τις εξαγωγές. Ευχαριστώ. Thank you. And the last coordinator present is Mrs. Ε, η κυρία Λέζινγκ είναι η τελευταία ε, συντονίστρια που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερωτήσεις ε, και οι ε, και οι των συναδέλφων νομίζω παρουσιάζουν το πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε αφενός ε, τα κριτήρια και την πραγματικότητα. Το θέμα λοιπόν το οποίο θέσατε κι εσείς είναι το πώς αυτά τα κριτήρια θα εφαρμοστούν καλύτερα ο κύριος ε, Φανόρντεν, ε, ε, αν κατάλαβα σωστά, αμφισβήτησε και τα κριτήρια τα ίδια. Είναι πράγματι μια πολιτική κατάσταση αυτή, δηλαδή εμείς καταλήγουμε σε κάποια κριτήρια, μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει πράγματι να τα ξαναδούμε. Ο κύριος Γκάλερ ξεκαθάρισε το πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή λέτε ναι, εντάξει, αυτά είναι αγκαία, αλλά υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αν υπάρχει κάποια σύγκρουση πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και μιλήσατε πράγματι για μια βιωσιμότητα. Κάτι το οποίο ε, κυριαρχεί στην Ατζέντα 2030. Μια βιωσιμότητα που δεν είναι μόνο οικολογική ο συνήθως, αλλά ε, νομίζω ότι εδώ πέρα σημαίνει ότι πρέπει από των προτέρων να πούμε το βήμα ένα ε, το οποίο κάνουμε, τι συνέπεια θα έχει στο βήμα 2, 3 και 4. Πολύ ε, πολύπλοκο αυτό, δηλαδή όταν μιλάμε για όπλα. Ποιος θα κρίνει κάτι τέτοιο, ποιος θα κρίνει π.χ. για την Γερμανία που εξάγει στη Σαουδική Αραβία σε βάθος χρόνου πολιτικά, οικονομικά, τι θα συμβεί και ποιος μπορεί να το εκτιμήσει. Ε, το θέσατε και εσείς κύριε Φανόρντεν. Δηλαδή μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και αλλιώς αυτό το ερώτημα. Εσείς λέτε ποιος από εμά ξέρει τελικά εάν χρησιμεύσαν σε κάτι όλα αυτά. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ ε, το ερώτημα εκ των προτέρων. Ε, ποιος από εμά ξέρει πόσο βλαπτικά είναι αυτά τα προϊόντα. Μιλάμε για φωνικά προϊόντα. Έτσι. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, κάνω σχόλια τώρα, αλλά ε, ε, οι συνάδελφοι έκαναν πολύ καλές ε, ερωτήσεις. Και νομίζω πως με αυτά τα οποία είπατε φάνηκε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της πολιτικής βούλησης και των πολιτικών αποφάσεων. Εκεί ειδικά όπου είπατε οι χώρες ε, όπως η Γερμανία και η Γαλλία δίνουν τα λιγότερα δεδομένα και μπορεί να είναι ζήτημα τεχνικών δυνατοτήτων. Ε, λίγο περίεργο όμως οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς να έχουν και τις λιγότερες τεχνικές δυνατότητες να δώσουν στοιχεία. Μάλλον παράλογο. Οπότε είναι νομίζω φανερά ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι σε ποιο βαθμό θεωρείτε εσείς ότι τελικά το πολιτικό επίπεδο είναι το επίπεδο το οποίο πρέπει να επηρεάσουμε. Έχουμε πολύ λεπτομερείς επιστημονικούς κανόνες και μια πρακτική για την οποία ε, υπάρχει αίσθηση ότι ό,τι και να λέμε δεν την αγγίζει τίποτα. Ε, Βεβαίω, εντάξει, γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορέ στα κράτη-μέλη. Μετά το ερώτημά μου το άλλο αφορά το κριτήριο 8. Είπατε πως είναι κάτι το πάρα πολύ ε, διαφορετικός προς την ερμηνεία του, επειδή έχετε πολλές ερμηνείες και είναι και επίμαχο, δηλαδή δεν είναι μόνο ζήτημα ερμηνείας, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν εντελώς. Και όταν τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας και της αναπτυξιακής πολιτικής και συνδέεται όλο και πιο στενά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κριτήριο Δηλαδή μια ακριβέστερη ερμηνεία αυτού του κριτηρίου και τελειώνω να επανέρχομαι στην Ατζέντα 2030 και το ερώτημά μου προς εσάς είναι αν έχετε την εντύπωση ότι οι θετικές εξελίξεις ε, στην Ατζέντα 2030 ε, πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση κοινωνικής ε, δικαιοσύνης και ειρήνης σε πολλές χώρες αν αυτό παραδείγματο χάρη επισέρχεται στον ορισμό και την αποδοχή του κριτηρίου 8. Γιατί τελικά το ζήτημα αυτό δεν θα έπρεπε να ερμηνεύεται τόσο διαφορετικά. αυτή είναι η προσωπική μου ερμηνεία, ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης Εντάξει, υπηρεσίες, υπηρεσίες, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάνε, ερμηνεύουν κτλ. Και στην πράξη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα συμβιβαστούν αυτά. Ευχαριστώ. Κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εδώ, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, σε πολλούς άλλους τομείς, έχουμε από τη μία τα κριτήρια και την διοντολογία και από την άλλη την πρακτική. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε για υποκρισία, νομίζω. Καταρχάς, με βάση τα κριτήρια που έχουμε, δεν θα έπρεπε να εξάγουμε σε χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ε, που είτε επιτίθενται, είτε υπάρχουν διάφορες ε, αντιμαχόμενες φράξεις. Παραδείγματο χάρη στο δημοκρατικό καθεστώ α πούμε τη Σαουδική Αραβία ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και όμω επειδή θεωρούνται φίλοι μα, εξάγουμε. Επομένω δεν εξετάζουμε αν η συμπεριφορά του είναι ε, εγκληματική ή όχι, αλλά αν η εγκληματική συμπεριφορά γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο ε, αποδοχής ε, από τους φίλους λοιπά, Ακόμα και αν ε, μαζικά, ας πούμε, αφανίζουν πληθυσμούς. Άρα έχουμε ε, δολοφονημένους δεύτερης κατηγορίας και εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Κίνα και η Ρωσία είναι οι κακοί, εμείς είμαστε οι κακοί. Ε, χρησιμοποιούμε βέβαια δημοκρατικές κορώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπερβολική ας πούμε, ευαισθησία όταν βλέπουμε τον βομβαρδισμό νοσοκομείων και τα παιδιά τα οποία αργοπεθαίνουν. Στην τηλεόραση βέβαια. Αυτά συχνά γίνονται, αυτές οι επιθέσεις γίνονται, θανατηφόρες επιθέσεις με όπλα τα οποία εξάγονται από την Ευρώπη. Και δεν μιλάω μόνο για την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει τεράστια ευθύνη, αλλά και για την Ισπανία που έχει μια σύμβαση με την ε, Σαουδική Αραβία, ε, Σαουδική Αραβία το οποίο σημαίνει ότι τα ναυπηγεία του Κάντιθ, τα οποία αργοπέθαιναν, θα μπορέσουν να πάρουν ε, έτσι μια ανάπαυλα ζωή, ας πούμε, ε, χάρη σε αυτές τις εξαγωγές ε, της Ισπανίας προς τη Σαουδική Αραβία. Από τη μία έχουμε τη ρητορία λοιπόν και από την άλλη έχουμε την, απρέξ, την απρέπεια. Και τι είναι στο μέσον, είναι η πράξη, ο ρεαλισμός, η realpolitik, η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι θετικό να κάνουμε, μια ε, να κάνουμε προσπάθεια να πλησιάσουμε την διοντολογία με την πρακτική. Αλλά τι γίνεται με τις εθνικές ανάγκες. Και μπροστά σε αυτές τα κριτήρια εξαφανίζονται και εμφανίζεται η σκληρή ανάλγητη πραγματικότητα. Από τη μία λοιπόν θα ήθελα να προσπαθήσουμε όχι να μιλήσουμε για την Κίνα ή για τη Ρωσία, να μιλήσουμε για τα δικά μα και για το πώ θα μπορούσαμε να παντρέψουμε πούμε, από τη διοντολογία με την πράξη, για να μην αποκλείουν τόσο πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριο Κέλαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τη Σίμπιλ εδώ, που θεωρείται πολύ αξιόλογη και σημαντική. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι χαρακτηριστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Απλώς ε, ο τομέας εδώ που μιλάμε είναι πιο ευαίσθητος. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους κανόνες και στην εφαρμογή τους. Οι ιδέες από τη μία και η πραγματικότητα, οι στόχοι, οι ανάγκες από την άλλη. Φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε από τη μία τις εθνικές, τους εθνικούς κλάδους, ας πούμε, ε, αμυντικής βιομηχανίας ε, που δεν έχουν και πολλή όρεξη να δώσουν πληροφορίες. Ας δούμε όμως καταρχάς ε, τις διαφορές ανάμεσα τις πληροφορίες που παρέχονται από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το διάλογο στα πλαίσια της ΚΟΑΡΜ. Επίσης, όπως είπατε, είναι σημαντικό το πόσο γρήγορα και το πόσο λεπτομερώς είναι αυτές οι εκθέσεις, το πόσο γρήγορα ε, εκδίδονται αυτές οι εκθέσεις αμέσως μετά ε, τις παραδόσεις. Γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες επίσης. Επίσης υπάρχει και αυτή η εργαλειοθήκη ε, μετά την επιβολή εμπάργου. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους. Ε, πώς μπορούμε εδώ να εμπλέξουμε και τις τρίτες χώρες. Πώς έχει η κατάσταση. Τα έχουμε καταφέρει, τις έχουμε εμπλέξει. Ο κύριος Γκάλερ ανέφερε επίσης ότι χρειαζόμαστε κοινέ πολιτικές. Καταρχάς σε επίπεδο χωρών. Εάν είχαμε κοινέ πολιτικές, τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουμε και την κοινή θέση σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων. Φυσικά, υπάρχει ένα δίλημα. Έτσι, πάντα. Ότι κάθε έθνος έχει δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του και να ζητήσει αμυντικά όπλα. Απ' τη μία, είμαστε πολύ απαιτητικοί από τον εαυτό μας και από την άλλη, προφανώς η Ουκρανία, ας πούμε, χρειάζεται αμυντικά όπλα. Και, αλλά κανένας δεν τις έδωσε. Και αυτό που αναφέρθηκε για τους μεγάλους εξαγωγείς όπλων, όπως η Κίνα και η Ρωσία, που δεν είναι τμήμα αυτού του συστήματος. Και νομίζω ότι αυτή η διαφορά, εμείς εντός του συστήματος και αυτή εκτός, έχει καταστροφικές ε, επιπτώσεις και για τη συμπεριφορά των ε, Ευρωπαίων εξαγωγείων όπλων. Ακούσατε κυρία μου λοιπόν πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις και σχόλια. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσετε αν έχετε σχόλια ή να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Με την ησυχία σας λοιπόν μπορείτε να απαντήσετε. Uh, και αν χρειαστεί θα επιτρέψω και δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Thank you very much. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Όλους σας πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και αφορούν μεγάλη ποικιλία θεμάτων για να τις δούμε μία-μία. Και αν θέλετε κάντε και επερώτηση για περισσότερες διευκρινήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις και το τι ακολούθησε το σύστημα διοδές των κρατών μετά την Αραβική Άνοιξη. Αν θέλετε ε, μία και μόνο απάντηση ότι θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους ε, εντελεχής αξιολόγηση. Έχουμε 28 διαφορετικές αποφάσεις αδειοδότησης, διαφορετικά συστήματα εξαγωγών από όλες αυτές τις χώρες, το δική του πρακτική και επίσης υπάρχει μεταβλητή της χώρας προορισμού. Άρα θα πρέπει να γίνει μια εντελεχής έρευνα στον background. Τι να σας πω, η απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνο με συστηματική ανάλυση τι μεταβολές έγιναν στους προμηθευτές αναχώρα. Άρα θα πρέπει να τα πω με τους συναδέλφους μου και να επανέλθουμε. Οι διαφορές τώρα αναπροορισμό ε, είναι κάτι το αυτονόητο να συγκρίνεται Λιβύη με Σαουδική Αραβία. Στη Λιβύη μπορεί να δείτε μεγάλη αλλαγή, μεγάλη πτώση, πάρα πολλές εξαγωγές όταν ήρθε το εμπάργο το 2003 2004 και υπήρχαν πάρα πολλά deal, πάρα πολλά ευρωπαϊκά όπλα. Βέβαια δεν έγιναν τόσες παραδόσεις παρά τα deal και μετά άλλαξε εντυπωσιακά η πολιτική αδειοδότηση. Άλλως έχουν τα πράγματα στη Σαουδική Αραβία, έχουν πάρει εκεί πάρα πολλά ευρωπαϊκά όπλα με διάφορες ε, αιτίες. Το θέμα είναι πολύ επίμαχο στα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν βέβαια αμυντικά συμφέροντα, υπάρχουν πολύ βαριά συμβόλαια, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και θέματα άμυνας, ε, μιλάμε για χώρες ήλους, οπότε θα πρέπει να τους δώσει κανείς, ε, να τους προσφέρει κανείς συνεργασία, οπότε αλλάζει έτσι η πολιτική. Άρα βλέπετε ότι είναι πάρα πολλά τα κριτήρια που επηρεάζουν την λήψη απόφασης. Γι' αυτό και είναι και σημαντικό να υπάρχει τελικά διαφάνεια για το πού καταλήγουν όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το κριτήριο, 8 ή αυτά τα 8 κριτήρια τέλος πάντων. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απόφαση για όταν θα δοθεί η άδεια. Αλλιώς είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει να κάνει με αυτή τη διαδικασία διοδότησης για το τι κριτήρια χρησιμοποιούνται. Άρα είναι περισσότερο θέμα διαδικασίας και όχι στην περίπτωση απόρριψης της ε, αίτηση τι γίνεται. Για το να κάνουμε τη μαύρη λίστα για το ποιος δεν υποβαλεί αναφορές. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει αξιολόγηση πιο εξισορροπημένη. Δεν είναι το θέμα ποιο ε, αναφέρει, ποιο αναφέρει, γιατί πολλέ χώρε υποβάλλουν ε, εκθέσει, αλλά ε, άλλο λέει για το τι άδειε δίνονται, άλλο για τι ποσότητε, άλλο για εξαγωγέ, άλλοι δίνουν περισσότερε πληροφορίε για του τελικού χρήστε. Άρα δεν είναι εύκολο να πει κανεί ποιο λέει πολλά, ποιο λέει λίγα. Και υπάρχουν και διαφορετικοί μηχανισμοί υποβολή αναφορών άλλοι υποβάλλουν στο, στον οργανισμό των συμβατικών όπλων. Άρα και εν προκειμένου θα πρέπει κανείς να κοιτάξει την κάθε χώρα προσωπικά για να είναι δίκαιος. Και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να πιέσουν την κυβέρνηση για ε, περισσότερες πληροφορίες αν κρίνουν ότι δεν αρκεί. Α, και το Ισπανικό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο. Γιατί πέρασε ένα νόμο που λέει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναφέρεται στην Κοινοβουλική Επιτροπή και το Αρμόδιο Υπουργείο. Άρα το Κοινοβούλιο δεν μπορεί μόνο να ζητεί πράγματα, αλλά μπορεί να ε, νομοθετήσει. Άρα ήταν πολύ δυναμικό σε αυτό το μέτωπο το Ισπανικό Κοινοβούλιο τώρα. Για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αυτό επίσης πρέπει να το αντικείμενο μελέτης. Ούτε αυτό προκύπτει από τις εθνικές εκθέσεις. Πρέπει κανείς να εξετάσει την κυβερνητική πολιτική, θα πρέπει κανείς να εξετάσει τα εθνικά κριτήρια που πολλές φορές έχουν να συμπληρώσουν τα οκτώ. Γερμανία, Σουηδία και άλλοι έχουν επιπλέον κριτήρια που σωρεύονται σε αυτά που προβλέπουν τα οκτώ. Οπότε πολλές φορές ε, υπάρχει το κριτήριο αυτών των δικαιωμάτων όπως στη Σουηδία. Το ίδιο και η Νορβηγία. Δεν έχει ως κριτήριο το ποιο είναι το όπλο, αλλά το ποιος είναι ο προορισμός της εξαγωγής. Επίσης, για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εξεταστεί και η συνθήκη ATT. Από το 2014 υπάρχει αυτή η Εθνή Συνθήκη για το εμπόριο των όπλων, οπότε οι πολιτικοί καλύπτονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήριο, οπότε δεν υπάρχουν μόνο τα ενωσιακά κριτήρια και τα εθνικά, αλλά έχουμε και αυτά τα δεσμευτικά διεθνή. Αυτό είναι μια νέα μεταβλητή που δεν υπήρχε όταν είχαμε το 1998 και την κοινή θέση του 2008 οπότε εδώ άλλαξε το σκηνικό και είχαμε διπλωματικές παρεμβάσεις από παντού διεθνώς. Κύριε Γκάλε, ρωτήσατε κάτι για τα εμπάργκο για τις διαφορές μεταξύ των εθνικών πολιτικών και την αξιολόγηση κινδύνου. Είναι σαφής η κατάσταση για ένα εμπάργο. Πρόκειται για απόφαση του ΟΗΕ ή καμιά φορά έχουμε και εμπάργο τη ΕΕ επί τη βάση κάποιας πολιτική εκτίμησης, κοινή. Και έτσι κρίνεται η τύχη των αδειοδοτήσεων. Αποτελούν κοινέ πολιτικές όσο υπάρχουν. Έχουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιστορικές σχέσεις χωρών με αποδέκτες και κατόπιν των εκλογών αλλάζει και η κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε ομοιογένεια στις αποφάσεις της αδειοδότησης ή στην ερμηνεία των ε, κριτηρίων ανταλλαγές απόψεων, διαβουλεύσεις, αυτά οδηγούν προς περισσότερη συνοχή της πολιτικής. Άλλος ρώτησε για το κατά πόσο έχουμε στοιχεία. Α, εσείς κύριε Αν έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα από τους ελέγχους των εξαγωγών. Αυτό είναι δύσκολο θέμα γιατί αν κανείς αποτρέψει κάτι, πώς θα αποδείξει ότι θα γινόταν, ότι θα συνέβαινε. Αυτό πάντοτε ισχύει με την αποτροπή των συγκρούσεων. Οπότε, εάν έχουμε παράδοση όπλων, στη συνέχεια έχουμε κάποια τραγωδία κατά πάση των δικαιωμάτων, αλλά τότε κανείς συνειδητοποιεί το ότι θα ήταν ποιο ήταν το συμφέρον κάποιο κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίθετο. Κάτι λέει ο κ. Βανόρντεν εκτό μικροφώνου. Είναι πολλέ χώρες που μπορεί κανείς να αναφέρει σχετικά. Αν ανατρέξουμε στην αρχή που θεσπίστηκαν τα οκτώ κριτήρια. Ε, αν δώσει κανεί όπλα σε αυτόν που θα αντιμετωπίσει αργότερα, είναι αυτονόητο ότι θα γίνει και γι' αυτό και είχαμε πολλές φορές και απόκληση απόψε, όπως με την Λιβύη. Τι έγινε με τα όπλα και ε, επίση στο Μαλί με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν όπλα εναντίον αυτού που τα είχε προμηθεύσει ή των συμμάχων του. Είναι θέμα ηθικής της πολιτικής, είναι θέμα χάρης που κάνει η Ένωση. Μα γι' αυτό και έχουμε αυτά τα κριτήρια, γιατί ε, είναι και θέμα του τι συμφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνει και τι να μην κάνει. Αλλά περάσαμε τώρα σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό ο σαν συνασπισμό κρατών. Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκέ λοιπέ χώρε. Και αυτή η συνθήκη ATT είναι πολύ κοντά. Συμπληρώνει την κοινή θέση που πάντα αφορά τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι, είναι ευρύτερη τη κοινή θέση η συνθήκη ATT. Έχει προσυπογράψει η Αμερική, αλλά η Κίνα και η Ρωσία όχι, γίνονται προσπάθειες να, να μπουν στη συνθήκη. Έχουν έρθει σαν παρατηρητές μια διαφορά οπότε ε, πολλές χώρε βέβαια συζητούν ε, τη συνθήκη ATT ότι είναι ένα όνειρο. Πάντως, εάν θέλετε περισσότερα στοιχεία για το πού οδήγησε το εμπόριο των όπλων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα πάτησή του να σας στείλω τέτοια στοιχεία για να δείτε τις λεπτομέρειες. Και εκεί λοιπόν πρέπει κανείς να κινηθεί περιπτωσιολογικά. Πάντως αυτό το επιχείρημα έχει γίνει βρέως. Επίσης, από το, την άξιση της γραφειοκρατίας, για το αν είναι κατόρθωμα να έχουμε πολυσέλιδες άδειες, ναι, είναι, γιατί θυμάμαι ότι παλιότερα οι εξαγωγές ήταν κάτι που γινόταν εν κρυπτό. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε γιατί ήταν λεπτό θέμα. Όμως βήμα-βήμα κατάλαβαν οι κυβερνήσει ότι θα έπρεπε τα πράγματα να γίνονται με λιγότερη μυστικότητα. Γιατί η μυστικότητα καλύπτει σκάνδαλα που είχαμε σε πολλές χώρες. Γερμανία, Σουηδία, Αγγλία. Και η μυστικότητα βοηθούσε τα σκάνδαλα. Και αυτή η εξέλιξη όσον αφορά τη διαφάνεια αντικατοπτρίζεται και στο τώρα απαιτούνται αυτές οι εκθέσεις των κρατών. Η κοινή θέση. Μεγάλη στροφή έγινε στο θέμα. από μία εικοσαετία το βασικό ήταν ότι είναι κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο, οι εξαγωγές, δεν επιδέχεται άλλη ανάλυση. Και αν θέλει κανείς πληροφορίες μπορεί να τις βρει από τη βιομηχανία. Δεν τους νοιάζει η μυστικότητα. Κάνουν το deal, δεν τους νοιάζει να το δημοσιεύσουν. Το μόνο το οποίο κρύβουν είναι η τιμή. Άρα μέχρι ότου συναυθεί η σύμβαση και η τελική τιμή, μέχρι τότε ενδιαφέρονται για μυστικότητα. Και έχουν το Συνταγματικό Δεστήριο στην ε, Γερμανία, με είχαν καλέσει ως εμπειρογνώμονα και εκεί οι δικαστές ρώτησαν τους εκπροσώπους της γεωμηχανίας να μπουν εντελεχώς τι γίνεται για το κάθε στοιχείο. Ποια σημεία, ποια στοιχεία και μέχρι πότε διέπονται από μυστικότητα και ακριβώς προέκυψε ότι ήταν το θέμα του πότε θα συνανθεί η σύμβαση και η τιμή. Και η σχετική απόφαση, όλα αυτά τα έγραφε και ονόματα των σχετικών εταιριών και όλα αυτά πήγανε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα πριν, υπάρχουμε, υπάρχουν πολλά αντιμαχόμενα αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Οπότε κανείς για να έχει ένα συμπέρασμα τεκμηριωμένο θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση και να πει έχω όλα αυτά τα δεδομένα και κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Και βέβαια δεν θα βρει το συμπέρασμα ο όλους σύμφωνος, αλλά τουλάχιστον θα έχει γίνει συζήτηση σε ένα κοινοβούλιο. Για να δούμε τώρα το άλλο θέμα. Τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και εδώ έχει οριμάσει προβληματική και στα πλαίσια του ΟΗΕ και για τη συνθήκη ATT και μου φάνηκε ότι είναι ενδιαφέρον το ότι ο πρόεδρος της διάσκεψης των χωρών συζήτησαν επί μέρες για τη σχέση μεταξύ συνθήκης για τα όπλα, ATT και βιώσιμης ανάπτυξης και είχαμε από τις ε, χώρες που συμμετέσχουν από Αφρική, Ασία, από όλες τις Υπήρους πολύ ευμενή σχόλια και υπήρχαν ε, ενδείξεις ότι υπάρχει σχέση ανάπτυξης και ελέγχου των εξαγωγών. Άρα εδώ συμφώνησαν και οι της ασφάλειας και της οι ασχολούμενοι με την ανάπτυξη. Και θα γίνει ακόμα μια διάσκεψη τον Σεπτέμβριο, οπότε και εκεί θα συζητηθεί το θέμα της ανάπτυξης. Επίσης, μας είπατε για Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία που έχουν δημοσιεύσει λιγότερες πληροφορίες. Μιλάμε όμως για παραδόσεις που έγιναν πραγματικά. Πάντως ε, όσον αφορά τουλάχιστον Γερμανία και Αγγλία υπάρχουν πολλά στοιχεία στι εκθέσει. Αν κάτσετε και τα με εκθέσεις άλλων, έχουν πει πολλέ λεπτομέρειες όσον αφορά αδειοδοτήσει. Αυτό αφορά και την Αγγλία. Είναι θέμα καλή πρακτική και έχουμε μελέτες για χώρες αποδέκτες και που εκεί αναλύονται οι πολιτικές των χωρών αποδεκτών που είναι πολύ ενδιαφέρον όταν περιλαμβάνεται σε μια τέτοια έκθεση. αυτό αυτόν αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, το κριτήριο 8. Το συζητήσαμε. Για να δούμε το επόμενο. Το επόμενο τι ήταν, οι παραδόσεις σε φιλικές χώρες και η συνοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά της δημοκρατίας. Σας παραμένω σε κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει στην Νορβηγία και ας μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ευθυγραμμίστηκε με την κοινή θέση. Αλλά και στη Σουηδία. ετήσει των κοινοβουλίων ζητήθηκε να διαπιστωθεί κατά πόσον η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τις ε, αδειοδοτήσεις προς μη δημοκρατικές, προς αυταρχικές χώρες. Άρα να μπει σαν κριτήριο στην αδειοδότηση το αν η χώρα είναι δημοκρατική. Αυτό ακόμα συζητήκεται σε Νορβηγία και Σουηδία, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προβληματική. Δεν είναι εύκολο να δοθεί ορισμός ποιο καθεστώς χαρακτηρίζεται αυταρχικό και πιο δημοκρατικό. Χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια, κάτι το οποίο όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά βέβαια είναι πολύ σημαντικό και για τις χώρες που αναφέρατε η Εμένη, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία, να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στο πλαίσιο της ε, άδεια εξαγωγής όφλων Και αυτό προξενή εντύπωση καμία φορά. Τώρα δεν θα αναφέρω χώρες. Δεν είναι σωστό να το κάνει το ΣΥΠΡΙ, αλλά μιλάμε για κράτη-μέλη της Ένωσης, όπου βλέπουμε ότι διαβολεύονται ελάχιστα με τα τμήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Υπουργείων. Δηλαδή, δεν φαίνεται να σχετίζονται τα ζητήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο να γίνεται με τρόπο συνεπή γιατί και πάλι στις ε, συζητήσεις για τη συνθήκη όπλων η Ένωση έχει κάνει πολύ σημαντικές δηλώσεις και ζητάει από άλλα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν. αυτό βεβαίως ενισχύει την εντύπωση ότι δεν είσαι και πολύ αξιόπιστος. Και γιατί βεβαίως ε, λέμε γιατί δεν μπαίνει η Ρωσία, η Κίνα κτλ. Και από την άλλη αν δεν έχουμε ενιαία εφαρμογή δεν βοηθάει και πολύ. Και θα αναφερθώ στην υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ακριβώς ε, το επίδικο ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση παραβίασε την σχετική συνθήκη. Αλλά δεν είναι εθνική η ευρωπαϊκή συζήτηση μόνο, αλλά χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης ε, που το σκέφτονται και λένε εντάξει καλά τα λένε οι Ευρωπαίοι θα το δουν αυτό το ζήτημα και οπωσδήποτε θα απασχολήσει τις διεθνείς συζητήσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και από τις γειτονικέ χώρες. Οπωσδήποτε νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκα σε κάποια από τα ζητήματα για το τι θεωρείτε ευαίσθητο από πλευράς πληροφοριών και είχατε και ακριβώ το θέμα του, ε, της εργαλειοθήκης για μετά το εμπάργκο. Το θέμα είναι βέβαιως πως υπήρχαν πολλές ε, ακριβώς ε, αρνήσεις, απορρίψεις, αλλά ελάχιστες πληροφορίες. Ε, Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο για το πώς αξιολογούνται κάποιες πληροφορίε ε, και πώς ερμηνεύουμε τα καρτήρια από του ανθρώπου που κάνουν αυτή τη δουλειά σε πραγματικό χρόνο, όχι ένα ή δύο χρόνια μετά. Ε, βεβαίω ε, η εργαλειοθήκη για μετά το εμπάργο είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Και αυτή ήταν η απόφαση, γιατί βεβαίω αν αρθεί το εμπάργο σε μια χώρα, Ακριβώς πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση αν θα πρέπει να τους δώσουμε όπλα αν μπορούμε να περιμένουμε, μήπως πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Και με τη Λιβύη, όπου πολύ ακριβώς ε, και Βεβαίω το ζήτημα της ανταλλαγής ε, πολιτικής σε σχέση με αυτή την χώρα. Αυτό μπορεί να επεκταθεί, να είναι πιο συχνές οι ανταλλαγές. Ε. Και το ιδεώδες θα ήταν βεβαίως ε, να μιλήσουμε για μια χώρα επίμαχη, επίχει η Σαουδική Αραβία. Για να γίνουν αυτές οι Ανταλλαγές δηλαδή. Να πούμε ναι, τώρα έχουμε διαφορετικές αξιολογήσεις, να τα συζητήσουμε λοιπόν. Οπότε τουλάχιστον να γίνει ένας διάλογος. έτσι ώστε κάποιες χώρες ε, να αλλάξουν τις θέσεις τους ε, κτλ. Για Ρωσία, Κίνα, ναι όπως είπα, είναι σημαντικός ο διάλογος με άλλες ε, χώρες και βεβαίως η συνθήκη εκεί νομίζω ε, είναι η κατάλληλη συνθήκη ελεγχόπλων, ναι, εμπορίου όπλων. Και πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ένα τέτοιο φόρουμ και με το ATT ε υπάρχει ακριβώς ε, αυτό το φόρουμ για πρώτη φορά και οι ευρωπαϊκές χώρες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, παρέχουν υποψηφίους για την Προεδρία, για τη γραμματεία, δίνουν λεφτά για το ταμείο, οπότε είναι ε, σχεδόν ευρωπαϊκή υπόθεση. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Αν όχι, παρακαλώ, ρωτήστε με. Υπάρχουν άλλες αρετήσεις. Κυρία Λέζινγκ. Θα μιλήσω γερμανικά. Έχω μία ερώτηση για τους τελικούς ε, χρήστες των προϊόντων. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μιλήσαμε ήδη για το Ισλαμικό κράτος, για την παράδοση όπλων στους ε, Πεσμεργά, ε, όπου τελικά αποδείχτηκε ότι κατέληξαν στο Ισλαμικό κράτος. Έχετε κάποιες προτάσεις ή ιδέες για το πώς ε, το πρόβλημα αυτό του τελικού χρήστη μπορεί να βελτιωθεί, πως μπορούμε ίσως να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ή να έχουμε κάποιους κανόνες, ας πούμε. Παρακαλώ. Θα απαντήσω αμέσως. Ναι, πολύ καλή ερώτηση για τους τελικούς χρήστες. Αυτό είναι τμήμα της αξιολόγησης κινδύνου. Ποτέ δεν υπάρχει ε, μια εγγύηση 100% για τον τελικό χρήστη, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει αλλαγή στην πολιτική κατάσταση μιας χώρας. Μπορεί να υπάρχει αστάθεια, κλοπή κτλ. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια λογική αξιολόγηση και η κυβέρνηση πρέπει να πει ότι αυτόν τον κίνδυνο είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε. Ε, πάντα υπάρχει. Για να ενισχυθεί η πιθανότητα τα όπλα να μείνουν στον τελικό χρήστη που ε, θέλαμε και να μην καταλήξουν αλλού, βεβαίως υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούν να γίνουν και βεβαίως Όλα αυτά είναι δηλώσει, υπογραφές κτλ. που όλοι ξέρουμε ότι μπορούν να πλαστογραφηθούν ή να αλλάξουν άποψη, ενδιαφερόμενοι κτλ. Μία επιλογή θα ήταν να έχουμε αποτελεσματικές κυρώσεις εάν δεν γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις. Και αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό εάν είναι μια κοινή γινουν σεβαστες οι δεσμευσει και αυτο θα ειναι πολυ δέσμευση η εγχείρημα. Π.χ. η Σουηδία ε, εξάγει όπλα σε μια χώρα, η χώρα τα δίνει αλλού. Δημοσιοποιείται αυτό. Η Σουηδία μπορεί να πει εντάξει δεν θα σου ξαναπουλήσουμε όπλα σουηδικά γιατί δεν μπορούμε να συμπιστευτούμε. Εάν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, που στηρίζουμε τη Σουηδία ούτε εμείς πουλάμε ε, αυτό θα είναι νομίζω σοβαρό αποτρεπτικό μέσο. Υπάρχουν επίσης και τεχνικές λύσεις ε, που αφορούν ε, την χνηλάτιση και Ακριβώ ε, το πώς μπορούν να σημαδευτούν τα όπλα και η βιομηχανία εδώ πέρα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αναζητά τέτοιες λύσεις για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα όπλα μέχρι τον τελικό χρήστη και να είναι προφανές εάν κάτι έχει κλαπεί από αποθήκες λοιπά. Και βεβαίως αν τα όπλα καταλήξουν κάπου αλλού μπορούμε να τα χνηλατήσουμε, να ξέρουμε πώς κατέληξε στους χύψη αντάρτες ή τρομοκράτες ε, το όπλο. Και υπάρχει βεβαίως ε, και το νέο γερμανικό μέσω των ελέγχων ε, μετά την αποστολή. Ο Γκάμπριελ τότε ο αρμοδιος υπουργός το είχε εξαγγείλει και ξεκίνησε τους ελέγχους μετά την αποστολή, δηλαδή να υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που να πηγαίνουν στις ε, χώρες και να βλέπουν αν οι παραδόσεις και τα όπλα είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Νομίζω θα γίνει στο προσεχές μέλλον. Γιατί πρέπει να γραφτεί στη σύμβαση δεν μπορεί να γίνει κάτι αύριο αν δεν έχουμε ενημερώσει τη χώρα εκ των προτέρων ότι αν σου στείλω όπλα τον επόμενο μήνα πρέπει να υπογραφεί μια σχετική ε, σύμβαση γιατί βεβαίω είναι και θέμα ε, κυριαρχίας της άλλης χώρας. Οπότε νομίζω πως υπάρχουν ε, πολλά και διαφορετικά βήματα. Και ένα άλλο θέμα αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να δελεγούν περισσότερες πληροφορίες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά παραδείγματο χάρη τις διαδρομές παράκαμψης ε, ή τα πλαστά πιστοποιητικά. Αν μια χώρα ξέρει ότι είναι πιθανόν τα όπλα να καταλήξουν αλλού, ε, δίνει αυτή την πληροφορία με, στους άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Ανέφερα επίσης την ε, σημασία ακριβώς του να υπάρχουν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες για να υπάρχουν και συναντήσεις μεταξύ των αρχών επιβολής ε, του νόμου. Πάντα είναι ηρωνικό ήδη από την πλευρά των ε, ειδών διπλής χρήσης αλλά και των όπλων ότι η αδειοδότηση, ότι αν θέλουν παραδείγματος χάρη αρμόδιοι για αδειοδότηση και επιβολή να συζητήσουν, το καλύτερο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να γίνει, ξέρω εγώ, σε Ασία, Λατινική Αμερική, μέσω μιας διάσκεψης για την οικοδόμηση δυνατοτήτων, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν. Αν προταθεί λοιπόν κάτι τέτοιο στο μέλλον, ελπίζω να το στηρίξετε για να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρα Μπάουερ. Τελειώσαμε λοιπόν με το εργαστήριο αυτό. Και σας ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής για την πολύ, πολύτιμη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ. Please stay. Next point of the agenda is... Περιμένετε για να ακούσετε το επόμενο θέμα που έχουμε την δεύτερη συζήτηση όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Ladies and gentlemen, please be seated. Those of you who wouldn't like to participate. Παρακαλώ καθίστε. Όσοι θέλετε να ακούσετε το επόμενο θέμα. Αλλιώς φύγετε. επόμενο θέμα. Κυρία Βάουτμαν, με την έκθεση της έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας θα μας μιλήσει για τις εταιρείε ιδιωτικής ασφάλειας. Είναι η δεύτερη φορά που εξετάσουμε αυτή την έκθεση. Την πρώτη φορά την εξετάσαμε το Μάρτιο 9 του μηνός. Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών ήταν η 16η Μαρτίου και τώρα έχουμε τη δεύτερη εξέταση του σχεδίου. Είναι εδώ οι ισχυώδεις συζητητές ε, για την έκθεση αυτή και χωρίς περαιτέρω σχόλια δίνω το λόγο στην κυρία Βάουτερ μας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους που διάβασαν και πρότειναν τροπολογίες στην έκθεση. Συνολικά έχουμε 343 ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν για να ε, βελτιώσουν το κείμενο. Έχουμε λοιπόν 19 συμβιβαστικές τροπολογίες και χτες ε, είχαμε νομίζω μια πάρα πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα και νομίζω συμφωνήσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό συμβιβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους και οδησηγητές από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύ καλή συνεργασία και τη γραμματεία βεβαίως για τις πολύ καλές χτεσινές διαπραγματεύσεις. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο ε, τελικά συνεργάστηκαν όλες οι ομάδες είναι το ότι είμαστε όλοι πεπισμένοι πως υπάρχει ένα κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ε, διάφορες δραστηριότητες αυτών των εταιριών και είχαμε κάνει μια κλειστή, ε, είχαν προτείνει μια κλειστή λίστα, μια μαύρη λίστα, αλλά με έψαν οι συνάδελφοι να έχουμε μια ανοιχτή λίστα με τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Δηλαδή να έχουμε μια θετική και όχι αρνητική αντιμετώπιση των εταιρείων. Επίσης ζητάμε η ευθύνη των δράσεων των ιδιωτικών αυτών εταιρείων να είναι σαφής ε, με τους συμβασμούς, ο οποίους καταλήξαμε θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι αυτές οι εταιρείε δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον στρατό και αυτό νομίζω τονίστηκε και με τις ε, τροπολογίες. Ζητάμε λοιπόν από Κομισιόν και Συμβούλιο να επεξεργαστούν ε, περισσότερες προδιαγραφές του πότε, πώς και γιατί ε, χρησιμοποιείται μια τέτοια εταιρεία σε διάφορες αποστολές και ζητάμε ακριβώς ε, να υπάρχει μια ειδοποίηση όταν θα τεθούν ε, τέτοιες εταιρείε κάπου όταν θα αναλάβουν δράση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια έκθεση ιδίας ε, πρωτοβουλίας, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ καλή συνεργασία. Thank you. Uh, now the shadow rapporteur for EPP is Mrs. Κυρία Ανδρουκάινεν, Κάινεν είναι σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Βάουτμαντς για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Μαζί με τους, σκιώδεις, τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές, νομίζω ότι εντοπίσαμε τα βασικά θέματα για τις δραστηριότητε αυτών των ιδιωτικών εταιριών, ε, για το πώς θα επιτηρούνται και θα, θα παρακολουθούνται. Το πιο σημαντικό σημείο της έκθεσης είναι ότι δίνει σαφή κατεύθυνση για το πώς οι υπηρεσίες των ε, ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ρυθμίζονται. Υπάρχει ανάγκη ε, να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εναρμονίσουμε τα νομικά πρότυπα για τις ιδιωτικέ αυτές επιχειρήσεις, που είναι διαφορετικά στα διαφορετικά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα αυτών των ιδιωτικών επιχειρήσεων που πληρούν τα υψηλά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τμήμα του ρυθμιστικού πλαισίου και να χρησιμεύει για να δίδονται συμβόλαια σε αυτές τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις ασφάλειας ε, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες αυτών των ε, επιχειρήσεων να είναι επιμελητιακού ε, χαρακτήρα προς, ε, προστασία περιοχών και όχι μάχημες δυνάμεις. Από το ιστορικό φαίνεται ότι η υπεργολαβία τοπικών ε, ιδιωτικών επιχειρήσεων Ασφάλεια δημιουργεί προβλήματα λογοδοσίας ε, και διάφαση. Γιατί δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίε ποτέ για τους υπεργολάβους. Η νομική ευθύνη γίνεται κάτι το πολύ αόριστο και οδηγείται στην ατιμορρησία και στην καταστροφή της φήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν η κοινή θέση είναι ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να δίνουν σε υπεργολάβους υπηρεσίες, απλώς μπορούν να προσλαμβάνουν ε, επιτόπου κάποιο προσωπικό για γλωσσικούς λόγους και για να τους δώσει ας γνώση της περιοχής κτλ. Επίσης, ε, θα πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοδοσία της χώρας ε, που κάνει αυτές τις προσλήψεις, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η χρησιμοποίηση προσωπικού στη συγκεκριμένη χώρα μπορεί να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας, εφόσον όμως οι υπηρεσίες παραμένουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να παροτρύνουμε την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να αναλύσουν το θέμα και να προτείνουν το κατάλληλο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας. Χθε είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και της εισηγήτριάς μας ε, και καταλήξαμε σε 19 συμβιβαστικέ τροπολογίε. Υπάρχει όμως ε, ένα ερωτηματικό για το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι δεσμευτικό προς τις επιχείρησεις και σε ποιο βαθμό. Εγώ ως ΕΛΚ, ε, ως τμήμα του ΕΛΚ, θα έρθω σε επαφή με την ομάδα μου πριν καταλήξω σε οριστική θέση για το θέμα αυτό. Ο κ. Φρονζουλίκα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και σκιώδεις εισηγητέ για την συνεργασία τους ε, στο σημαντικότατο αυτό θέμα. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας στην Ευρώπη συνεχίζεται και αυξάνεται κάθε χρόνο. Και αν λάβουμε υπόψη το ότι δραστηριοποιούνται σε υπερεθνικό επίπεδο, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τεράστια προβλήματα ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λάβουμε ειδικά υπόψη ότι η ανεπαρκή διαφάνεια, η ανεπαρκή μηχανισμοί παρακολούθηση και η ανεπαρκή ε, λογοδοσία των επιχειρήσεων στα θέατρα επιχειρήσεων είναι προβληματική. Στη χθεσινή συνάντηση των σκιωδών εισηγητών χαίρομαι που φτάσαμε σε συνένεση σε, στις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες που πρότεινε η εισηγήτρια. Όμως, συνάδελφοι, όμως, να τονίσω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μία επισκόπηση, μία λεπτομερή αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης για αυτές τις ε, εταιρείε που έχουν έντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είτε δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε τρίτες χώρες και παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκούς ή μη ευρωπαϊκούς φορείς. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ρυθμιστικό μοντέλο, που μεταξύ άλλων θα εξασφαλίζει την αναφορά παρατυπιών, ε, παρανομιών από πλευρά αυτών των επιχειρήσεων και πλέον να λογοδοτούν, να μπορούν να λογοδοτούν οι επιχειρήσει αυτέ. Ε, το γεγονό ότι δεν είναι ομοιογενεί οι εθνικέ νομοθεσίε και κάποιε ρυθμίσει ε, που έχουν οι ίδιε οι επιχειρήσει ε, οδηγούν σε καταχρήσει και έχουν τεράστιε επιπτώσει στο πώ λειτουργούν σε πολυμερείς επιχειρήσεις οι εταιρείε αυτές και σε συγκρούσεις, σε περιοχές και χώρε συγκρούσεων. Επίσης, εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις ε, επιχειρήσεις για να υποστηρίξουμε τις ε, στρατιωτικέ και μη στρατιωτικέ ε, αποστολές μας και το προσωπικό μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η χρήση που κάνουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις καθορίζει και το πώς μας βλέπουν οι άλλοι και την εμπιστοσύνη που μας έχουν οι ιδιωτικέ επιχειρήσει μπορεί να παίξουν ε, σημαντικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατεία και στην ε, αύξηση της ασφάλειας της θάλασσας. Όμω, η δημιουργία ένοπλων ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλεια έχει δημιουργήσει ειδικά προβλήματα σε θαλάσσιο επίπεδο, γι' αυτό θα ήθελα ένα ειδικό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τη θάλασσα. Αυτά και σας εύχομαι και καλό Πάσχα. Ναι, ναι, έχουμε χρόνο για τις ευχές. Mr. Buchner for Ο κύριος Μπούχνερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με ναι, όλα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το έγγραφο το οποίο προέκυψε. Ένα πράγμα είναι σημαντικό και θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και καιρό στην Επιτροπή μας. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα οδηγήσει σε, κάποια, σε ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν γίνει αυτό τότε κάπου θα χάθει αυτή η υπόθεση. Αυτό έχω να πω εγώ λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια που δεν ζητάει κάποιος άλλος ε, τον λόγο, η κυρία Βάτμαν θέλει ξανά να μιλήσει. Η συγκέντρια σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ με όλους όσους έλαβαν το λόγο. Με, θα δω τις τροπολογίες, θα στείλω τις συμβαστικές του συναδέλφους και θα τα ξαναπούμε κατά την πράσινη εβδομάδα. Καλό Πάσχα και σας ευχαριστώ. Επίσης, επίσης, να πολύ καλό Πάσχα εύχεται και η Πρόεδρος. Συνάδελφες, στην Άφελ θα γίνει ψηφορία 2 ή 3 Μαΐου. Οπότε παρακαλώ όσοι συμμετέχετε εκεί να είσαστε παρόντες στην ΑΦΕΤ τότε για την έγκριση αυτής της έκθεσης. με αυτό το θέμα. Όποιος φύγει τώρα, του εύχομαι καλό Πάσχα, αλλά μείνετε παρακαλώ γιατί έχουμε το επόμενο σημείο με εξαιρετικές παρουσιάσεις. I think we uh, Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Περίπου πέντε λεπτά επομένως. Για ένα τσιγαράκι, ίσως.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

Colleagues, please be λέει ο Πρόεδρο. Ωραία. Πρόκειται για το τελευταίο σημείο της ημέρα τη δίδαξη. Τελευταίο, αλλά οπωσδήποτε πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την αναθεώρηση των δομών διαχείρισης Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρίσεων πολιτικού και στρατιωτικού συντονισμού. Και με μεγάλη μου χαρά εύχομαι το καλό όρισαν στους δύο προσκεκλημένους μας. Τον ένα τον γνωρίζετε και από χθε. Από τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε και είναι ο διευθυντή της CPCC, ο Κένεθ Ντίν, στα πλαίσια της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράση. Επίσης έχουμε και τον Πολωνό προσκεκλημένο μας, τον κύριο ε, υπονάβαρχο Βάλτεμαρ Γκλούσκο που είναι πληρωτή αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ορίσατε, κύριε, στην συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας. Έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει να παρουσιάσετε, οπότε και ευθύ αμέσω θα σα δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Κεναθντίν και στη συνέχεια στον υπονάβαρχο. Σας ευχαριστώ που με ξανακαλέσατε. Πάντοτε είναι πολύ ευχάριστο να έρχομαι εδώ. Και βεβαίω είναι θέμα του Βάλτεμαρ. Εκείνο έχει την κύριο συντολή. Αλλά εγώ από πλευράς ε, πολιτικού προσωπικού, από ε, πολιτικού σχεδιασμού να σας πω πώς το βλέπουμε. Άλλωστε έτσι ε, ονομάζεται και η υπηρεσία μας. Εδώ και μια δεκαετία ασχολούμεθα με αυτό το ζήτημα και έχουμε αντιλήσει σε αυτή τη δεκαετία κάποια συμπεράσματα, αλλά ακόμα μαθαίνουμε. Ακόμα προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Και άλλωστε και χθε τα συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να έχουν περισσότερη ετοιμότητα, περισσότερη αμεσότητα και για υποστήριξη αποστολών και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας. Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, πάντως λαμβάνοντας υπόψη και με σεβασμό τον ρόλο των στρατιωτικών συναδέλφων και έχουμε εδώ πέρα τα θέματα, τα ιατρικά, την υποστήριξη, τη μεταφορά, την υλικοτεχνική υποστήριξη και επιμελητία και οπότε εμείς από πλευράς ε, πολιτικού κλάδου αυτά τα θεωρούμε θετικές εξελίξεις. Έτσι παίρνει σάρκα και οστά και το δικό μας έργο. Πάντοτε στο θέατρο επιχειρήσεων όπως το Μαλί και στην Σομαλία. Εκεί πιάνουν τόπο αυτά. Έχουμε τους όλους τους εκπροσώπους και τις αντιπροσωπίες των Ευρωπαίων που βρίσκονται εκεί και τις αποστολές. Θα πρέπει επομένως συνεχώς να ασκούμε αυτοκριτική, να προσέχουμε τι κάνουμε, τι λέμε, ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαία θέση. Δεν εκπροσωπούμε τις χώρες μας, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς από πλευράς πολιτικού προσωπικού και υπάρχει και το θέμα του στρατιωτικού συντονισμού. Και βέβαια για την προσωπία μας φροντίζει τα πολιτικά και τα οικονομικά. Οπότε θα πρέπει έτσι να προβληματιζόμαστε για το πώς θα κάνουμε το καθήκον μας επί τη βάση της εντολής μας έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Και επομένως προχωρεί τη διαδρομή της η υπηρεσία μας, η CPCC, αλλά τώρα και με την υπηρεσία του Βάλτεμαρ συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει να έχουμε κοινό προγραμματισμό και κοινή ε, συμπεριφορά ούτως ή Όχι μόνο εδώ στις αλλά και στο θέατρο των επιχειρήσεων. και πάντοτε θα πρέπει να κινούμεθα στα πλαίσια του προπολογισμού της ΚΕΠΑ. Και όσο πιο πολύ καθιερώνεται ο ρόλος μας θα πρέπει να βλέπουμε και να προσπαθούμε στο θέατρο επιχειρήσεων να έχουμε ενιαία στάση και συνεργασία. και ενιαίο μέτωπο ούτως είπε. Σας βεβαιώνω ότι εμείς από πλευράς μη στρατιωτικής δυνατότητας σχεδιασμού κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βλέπουμε το στρατιωτικό σκέλος ως ανταγωνιστή. Για μας αποτελεί μια ικανοποίηση η συνεργασία με την υπηρεσία του Βάλτεμαρ όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι θα πρέπει να μας στείλει ως αποστολή. Ευχαριστώ. Και τώρα να πληρωτήσει αρχηγό του Στρατιωτικού Επιτελείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Καταρχά, θα ήθελα να ξεκινήσω εξηγώντα το λόγο για τον οποίο θέλουμε να προσαρμόσουμε τη δομή διαχείρισης των κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση στο γιατί, επίσης την απάντηση στο τι σκοπεύουμε να κάνουμε και στο πώς σκοπεύουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Καταρχάς, η πρώτη ερώτηση είναι το γιατί. για τις ε, μη εκτελεστικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα διάφορα επίπεδα διοίκησης, ξεκινώντας από το στρατηγικό ε, και πηγαίνοντας προς το τακτικό, όλες αυτές οι ευθύνες ε, τις είχε ο διοικητής της αποστολής επιτόπου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο διοικητής αυτός θα έπρεπε να πηγαινοέρχεται ε, από το αρχηγείο του στο Μαλί, στη Σομαλία και <laughs> να πηγαίνω έρχεται στις Βρυξέλλες. Είχαμε περιπτώσεις ε, που διακυβευόταν και η ακαιρεότητα της αποστολής. Όταν έλειπε, ας πούμε, ο διοικητής από τους στρατιώτες του. Στρατιωτικός, πώς αυτό είναι απαράδεκτο. Προσπαθούμε, λοιπόν, να δούμε σε στρατηγικό επίπεδο διοίκησης ε, τι μπορούμε να κάνουμε στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό οι ανακατατάξεις αυτές. Επιπλέον θέλουμε να υπάρχουν περισσότερε συνέργειες ανάμεσα στις ε, στρατιωτικές και μη στρατιωτικέ αποστολές. Γίνονται συζητήσεις εδώ και καιρό για το πώς μπορούμε να αλληλοϊποστηριχθούμε επί τόπου. Παραδείγματο χάρη στο Μαλί έχουμε μία και στρατιωτική και μη στρατιωτική αποστολή και οι δύο συνεργάζονται βεβαίω Αλλά σε ό,τι αφορά τις επίσημες, ε, τον επίσημο διακανονισμό, ας πούμε, τα πράγματα ήταν ασαφή και δύσκολα. Όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις δομές που προβλέπει. Σε ό,τι αφορά το τι, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου λένε ότι ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μόνιμη ε, δυνατότητα σχεδιασμού ε, για τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμεινο για του 2017. Μόνιμα καταρχάς, και αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα μέχρι τέλος ε, Ιουνίου, και μία απόφαση για να βασιστούμε στις δομές της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τα συμπράγματα του Συμβουλίου είχαν στις 6 Μαρτίου του 2017 είχαν ε, στοιχεία για το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Και είπαν ότι αυτές οι νέες δυνατότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ε, δυνατότητες ε, στρατιωτικού σχεδιασμού και θα πρέπει να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στη δομή ε, στρατιωτικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Διευθυντής του στρατιωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τα καθήκοντα και αυτό ήταν αποτέλεσμα μακράς πολιτικής συζήτησης, τελικά θα λέγεται διευθυντής του, των δυνατοτήτων σχεδιασμού, στην πράξη θα έχει καθήκοντα στρατιωτικού διοικητή. για τις δυνάμεις ε, που έχει στην, που υπάρχουν σε αυτό το, στο επίπεδο του, Και ο επιχειρησιακός διοικητής θα σχεδιάσει ποιος κάνει τις επιχειρήσεις και ποιος είναι υπεύθυνο για τις μη εκτελεστικές ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, μη επιχειρησιακές μάλλον επιχειρήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τρεις αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει και μια τέταρτη όμως, θα είναι επίσης δική του ευθύνη. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις ε, αρμοδιότητες για το Αθήνα, θα έχει το ρόλο του διατάκτη του προπολογισμού, στο ποιο είναι δηλαδή είναι υπεύθυνο για τα θέματα προπολογισμού, εκτέλεση του προπολογισμού κτλ. Όπω είπα επίση, σε ό,τι αφορά τι συνέργειε ανάμεσα στο ιδιωτικό και μη στρατιωτικό σκέλο, που προβλέπεται μέσω τη εφαρμογή αυτή τη νέα δομή, αναμένουμε να, να υπάρχει ένα πυρήνα συντονισμού για την αμοιβαία υποστήριξη ούτω ώστε να υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στι δυνατότητε ε, στρατιωτικού σχεδιασμού, σχεδιασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων και τι δυνατότητε σχεδιασμού μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ε, συζητάμε για το ποιο θα είναι σε αυτόν τον πυρήνα, πώ θα γίνεται ο συντονισμό, Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή όμω, χρειαζόμαστε χρόνο. Ε, είναι α πούμε μια διαδικασία. Έτσι. Και καταρχά για μας η προτεραιότητα είναι να έχουμε πρώτα δυνατότητε ε, σχεδιασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων Έχουμε ήδη εντοπίσει τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται. Και όταν είπαμε ότι το ελάχιστο δυναμικό του επιχειρήν έχει... το έχουμε φτάσει, αυτό σημαίνει ότι ο επικεφαλής, ο, δηλαδή ο διευθυντής της αποστολής, κάνει αυτό που πρέπει. Σε στρατιωτικό επίπεδο ε, έχουμε τον ΟΠΚΟΝ, που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, για την εφαρμογή του σχεδίου, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων και την προσαρμογή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων με βάση το, τις εξελίξεις επιτόπου. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία για τα οποία είναι υπεύθυνο. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Ο πυρήνας ε, αναζητάται από, το στρατιωτικό προσωπικό. Κάποιοι αξιωματικοί θα έχουν διπλή ιδιότητα. Θα κάνουν τη δουλειά τους εντός του στρατιωτικού, της στρατιωτικής διοίκησης και παράλληλα η γνώση τους θα χρησιμοποιηθεί και για τις αποστολές ή για την αποστολή. Όσοι επίσης είναι εξοικειωμένοι με τις επίσημες διευθετήσεις, τους επίσημους διακανονισμούς μέχρι τα τέλη του 2016, η οντότητα που λέγεται Activated Operated Center, Operation Center ε, απενεργοποιήθηκε, αλλά το προσωπικό μέσα σε αυτό το κέντρο και μετακινήθηκε και δημιουργήθηκε κάτι που ονομάζεται ενδιάμεση έντος, ε, οντότητα, που είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του MPPC. MPCC, συγγνώμη. Και μιλάμε για την οργάνωση, για τις ε, μόνιμες διαδικασίες ε, των επιχειρήσεων, μιλάμε για υποδομή, για περιγραφή των διαφόρων θέσεων, για όλο το προσωπικό που ασχολείται με το MPCC. Σε ό,τι αφορά την, ε, τις προδιαγραφές της κάθε θέσης, Μέχρι 31 Μαρτίου ήταν έτοιμε όλε αυτέ οι προδιαγραφέ ε, και υποβλήθηκαν προ σχολιασμό από τα κράτη-μέλη. Και τα τελευταία σχόλια ακούστηκαν χθε και τα κατέγραψε το στρατιωτικό προσωπικό. Θα ετοιμάσουμε το επόμενο σχέδιο μετά το Πάσχα, τρίτη μετά το Πάσχα, τρίτη του Πάσχα. Και μέχρι τις 28 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης, εξηγήσαμε στα κράτη-μέλη ότι περιμένουμε την εφαρμογή από μέρους τους για τις θέσεις ε, εντός του MPCC ε, με απλή ιδιότητα. Όλα είναι συμπιεσμένα χρονικά, όλα θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι τις 10 Ιουνίου, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Να βάλουμε το σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση καταρχάς και όλη η διαδικασία θα πρέπει να γίνει σύμμορφα με τους κανόνες. Περιμένουμε λοιπόν τις δύο-τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου. Θα πρέπει να συγκαλέσουμε δεκάδες ε, συμβούλια επιλογής προσωπικού, οι οποίες θα διεκπαιρεώσουν τις αιτήσει που θα εξετάσουν και διεκπαιρεώσουν τις αιτήσει που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη. Έχουμε και μία ενδιάμεση δυνατότητα επιχειρήσεων του MPCC, όπου ε, μέχρι τις 18 Μαΐου περιμένουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δημιουργία του MPCC και τις αποφάσεις του Συμβουλίου που αλλάζουν τις τρέχουσες αποφάσεις για τις μη εκτελεστικές ε, επιχειρήσεις, των τον διευθυντή δηλαδή, καταρχάς, του στρατιωτικού σχεδιασμού κτλ. σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Όλα τα διοικητικά έξοδα που συνδέονται με, τις, ε, με τα γραφεία, με τις υποδομές, ε, την πληροφορική, την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων, όλα θα, θα τα λάβουμε από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης. Σε ό,τι αφορά το κόστος αυτό καθεαυτό των επιχειρήσεων, κάποιες από αυτές έχουν δικαίωμα να αντλήσουν χρήματα από το κοινό ταμείο του Αθήνα. Τέλος. Όπως λένε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η λύση στο πρώτο βήμα, στο πρώτο επίπεδο, θα είναι κάτι που θα εφαρμοστεί πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αυτό το πρώτο, η πρώτη εφαρμογή δεν θα είναι τέλεια και προβλέπουν τα συμπέρασμα του Συμβουλίου ότι η MPCC ε, με αυτόν τον κοινό πυρήνα συντονισμού θα επανεξεταστεί ένα χρόνο μετά, μετά από τη δημιουργία του φορέα αυτού, του πυρήνα αυτού, όχι αργότερα όμως από το 2018. Αυτή είναι η φάση στην οποία έχουμε φτάσει τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις. Okay. Uh, I open. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γκάλερ. Τσιγκούιε Μπάρτσο Ναύαρχε. Και σας ευχαριστώ και κύριε Ντίν. Ενδιαφέρον το ότι μας φαίνεται και ευχάριστα για, τον, για την ίδρυση του NPCC, οπότε έχουμε τώρα ε, και το άλλο τμήμα του ζεύγους. Ε, το CPCC, το πολιτικό σκέλος υπήρχε, το NPCC βεβαίως αφορά τις μη εκτελεστικές αποστολές. Αλλά Τέλος χαιρόμαστε που σας έχουμε σας ως ειδικούς εκεί όπου ε, θα πρέπει να είστε και μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε ως Κοινοβούλιο να πιέσουμε εμείς ε, τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και ακριβώς ε, αυτό είναι χαρακτηριστικό όταν περιγράφει κανείς πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί ένα όνομα για τον διοικητή των επιχειρήσεων χωρίς να το πούμε, χωρίς να το πούμε διοικητή επιχειρήσεων. Ε, μα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή Ελπίζω να μην είναι η δικιά μου η χώρα που δημιουργεί τα προβλήματα, ελπίζω να είναι η χώρα η οποία αποχωρεί. Αλλά πρέπει ε, να σταματήσουν τώρα αυτές οι κολυσιεργίες. Αν κατάλαβα καλά, ο διοικητής ήταν αυτός ο οποίος θα εγκρίνει και τις δαπάνες ε, για την Αθηνά Νομίζω ότι είναι ένας ε, τομέας όπου εμείς ως ε, Κοινοβούλιο πάντα ήμασταν σαφείς. Καθώς θέλουμε να επεκταθεί το πεδίο της Αθηνάς, ε, να μπορούν τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν σε είδος, για να μετρήσει το κόστος έτσι ευρύτερα. Και άλλοι να συνεισφέρουν σε χρήμα και να μην εκστρατεύουν. Τέλος πάντων, πώς ε, έχουν οι συζητήσεις. Εσείς που ε, τα βλέπετε στην πράξη. Πώς βλέπετε την διαθεσιμότητα δυνάμεων. Θεωρείτε ότι θα είναι πιο εύκολη η κατάσταση αν επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή της Αθηνάς. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ όσων κάνουν αυτές τις αποστολές και πώς παρακολουθείτε την πολιτική συζήτηση. υπάρχει κάποια ελπίδα να επεκταθεί στο προσεχές μέλλον. Ίσως ε, θα μπορούσαμε, δεν ξέρω, να έχουμε μια απόφαση τον Ιούνιο για ενεργοποίηση. Ίσως έχουμε και άλλες ενθαρρυντικές αποφάσεις για την Αθήνα. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λέζινγκ. I would like to Θα μιλήσω γερμανικά. Έχω πρώτα απ' όλα μία ερώτηση στον κύριο δίν. Στην ε, συζήτηση για την κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας υπήρχαν κάποιοι που προειδοποιούσαν για την στενή διαπλοκή ε, στρατιωτικής και πολιτικής διαχείρισης κρίσεων. Θυμάμαι π.χ. το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ειρήνευσης. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Αυτή η διαπλοκή αλλάζει καθόλου ειδικά σε σχέση με τον πολιτικό τομέα όταν οι στρατιωτικές δομές εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων. Έχουμε ήδη εμπειρίες. Έχετε κάποια σχετική πείρα και αν ναι σε ποιο βαθμό. Μετά είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι στο Μαλί, παραδείγματο χάρη, ε, δίνεται το βάρος ε, σε μια ενιαία παρουσία της Ένωσης. Σημαίνει αυτό τελικά ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ της ε, πολιτικής επιχείρησης ε, και και των στρατιωτικών πτυχών. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις εμπειρίες του Αφγανιστάν, όπου είχαμε καλέσει διάφορες ΜΚΟ που μας είπανε ότι αυτό είναι μειονέκτημα γιατί δεν τους θεωρούν πλέον ε, μικιό ε, και μπορεί να υπάρχουν και πολεμικές επιχειρήσεις ακόμα και αν δεν θεωρείται μια επιχείρηση ως τέτοια. Π.χ. στο Αφγανιστάν ε, επιτέθηκαν κάποιοι στα αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού και δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Τι γνωρίζετε αυτούς τους ε, κινδύνους. Σας ε, ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για τους δύο, και τους δύο ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπαν. Και επίσης όλα αυτά είχαν αισιόδοξο τόνο. Αρκετά αισιόδοξο. επιτέλους βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά για να επανέλθω στα όσα συζητήσαμε στην αρχή. Δεν τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητούμε. Το θέμα επομένως δεν είναι μόνο ο συντονισμός. Σε επίπεδο υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Έχουμε κάποιες υπηρεσίες που κάνουν τον προγραμματισμό των αποστολών. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστή διαχείριση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ζήτημα αυτό που συζητούμε τώρα θα είναι βασική προτεραιότητα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Θα θεωρείται δηλαδή ανάγκη, αναγκαιότητα και όχι ε, πάρεργο ας πούμε παρεμπίπτους απασχόληση τέλος πάντων. Για τα άλλα τώρα. Έχω δίκιο να θεωρώ ότι οι περισσότερες λειτουργίες περί της αποστολές έχουν μεικτό χαρακτήρα πολιτικό και στρατιωτικό. Ε, αυτό θα πρέπει να μας κάνει υπερήφανος. Αν ισχύει αυτό που λέω. Ε, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της πολιτικής υπηρεσίας και ποιες της στρατιωτικής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει διαφορετική δομή, διαφορετική προϊστάμενη για κάθε κλάδο. Ακριβώς όμως Πώς ε, καθορίζεται η ιεραρχία μεταξύ τους ή όσον αφορά τον επικεφαλής ε, της κάθε φορά επιχείρησης. Ο κύριος Γκάλερ έδειξε κάποια ενδιαφέροντα το ζήτημα των ε, δυνατοτήτων, αλλά σήμερα μιλάμε για τις δομές διαχείρισης. Για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτές τις δομές διαχείρισης όμως, θα πρέπει να φροντίσουμε τις δυνατότητες και τις θετικές και τις πολιτικές. Δηλαδή, το ζουμί είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή δυνατότητα. Τέτοιου είδου επιχειρήσεις θέλουμε να έχουμε. Να αξιοποιούνται και να συνδυάζονται οι δυνατότητες όλων των κρατών μελών. Είναι βέβαια και θέμα του προϋπολογισμού των μελλοντικών προϋπολογισμών. Ξέρω ότι έχουν εγγραφεί κάποια κονδύλια ε, για την πολιτική ασφάλειας και τα σχετικά. Όμως, ας κάτσουμε να αναλογιστούμε. Τι μπορούμε να πετύχουμε παραπάνω, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπάνω από το τι κάνουν το κάθε κράτος μέλος χωριστά. Άρα, αυτό πρέπει να πει δυνατότητες που θέλουμε να προσδώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπίχνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μου δώσατε τον λόγο. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους δύο προλαλήσαντες. Πρέπει να πω ότι προσωπικά εγώ έχω δυσκολίες για το ότι έχουμε αυτή την ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Δηλαδή τα δύο πάνε μαζί. ε, κάπου πρέπει να συζητήσουμε ακριβώς ποιο είναι το όριο μεταξύ των δύο. Τέλος, αν θέλω να ρωτήσω. Ποιος δίνει τις διαταγές, ποια είναι η αλυσίδα της ιεραρχίας, πού είναι ο διαχωρισμός και πώς έχει η αλυσίδα της ιεραρχίας με την συνεισφορά του κάθε κράτους μέλους. Ε, μιλάω για τους στρατιώτες. Πώς ε, πηγαίνουν οι διαταγέ λοιπόν, ποια είναι η αλυσίδα τη ιεραρχία, Η πρόεδρος δεν ε, ζητεί άλλος το λόγο, αλλά θα ήθελα εγώ να υποβάλω ερώτηση σε σχέση με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Γιατί να έχουμε νέες δομές διαχείρισης, τι είδους είναι αυτές, πώς θα το καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Και έχω επομένω ε, μια γενικότερη ερώτηση, έτσι όπως πάντα να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή ότι θα πρέπει να μην έχουμε επικάλυψη ενεργειών με το ΝΑΤΟ. Πώς ακριβώς θα το αποφύγουμε αυτό. Πώς δεν θα έχουμε επικάλυψη επομένως με τις δομές και τα θέματα του ΝΑΤΟ. Έχετε το λόγο αγαπητοί με την ίδια σειρά. Πρώτα ο κύριος δίνεται και κατόπιν υπονάβαρχος του Γκλούσκου. Πρώτα πρώτα για την κυρία Λέζινγκ. Συγγνώμη αν κάτι δεν σας το είπα ξεκάθαρα. Ναι, έχω κάνει και στο Αφγανιστάν και καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διέρη και βασίλευε με τα διάφορα προγράμματα. Και η εμπειρία μου από το Αφγανιστάν ήταν ότι πολλές φορές ο κακός μπάτσος είναι στρατιωτική και το πολιτικό σκέλος είναι ο καλός ο μπάτσος. Γι' αυτό και πολλέ φορέ όπου είναι υπερτονισμένη η στρατιωτική πτυχή είναι αποφευκτέ κάποιε αποστολέ για κάποιου. Αποστολέ εκένωση κλπ. Οπότε αυτό το one entry μην το παρεξηγείτε. Θεωρώ είμαστε μία οικογένεια. Χρειάζεται συνέργεια. Αλλά υπάρχει χωριστή ιεραρχία. Η λειτουργία είναι παράλληλη και υπάρχουν χωριστές εντολές. σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει, υπάρχει κάποια πολιτική διέργεια βασίλευε Τώρα όταν λέμε για αναβαθμισμένη συνεργασία και συνέργειες, αυτό δεν αναιρεί τις χωριστές ιεραρχίες. το πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η ιεραρχία τι σημαίνει και έτσι θα οικοδομήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Ένα πούμε είμαι εγώ, ο επικεφαλής της επιχείρησης, εδώ στις ε, ε, Βρυξέλλες. Αλλά υπάρχει και κάποιος επικεφαλής που ασκεί τη διοίκηση στο θέατρο των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό Έχετε δίκιο κύριε Γκάλερ. Υπάρχει και θεωρητικός διοικητής. Δεν είναι θέμα το πώς τα λέμε. Ξέρετε γιατί χρησιμοποιείται αυτή την ορολογία. Πρόκειται για το διευθυντή της MPCC ε, και υπάρχει και ο άλλος της CPCC. Πώς να το εξηγήσουμε, δεν είναι εύκολο. Οπότε ο διευθυντής της έμπισης είναι ο επικεφαλής των επιχειρήσεων, ο οποίος αναφέρεται στον διευθυντή της υπηρεσίας εδώ, όπως και εγώ. Και αυτά επί τη βάση της κτηθήσης εμπειρίας. Θα σας τα εξηγήσει και ο Βάλτεμαρ για το πώς το στοιχειωτικό σκέλος λειτουργεί. Γιατί είναι σημαντικό στοιχείο η ιεραρχία. Να μην επεμβαίνει το στοιχειωτικό σκέλος στο πολιτικό. Υπάρχει επομένως διαχωρισμός όσον αφορά την στοιχειωτική δομή. Αλλά για ασφάλεια, για επικοινωνίες, για υποστήριξη λιγοτεχνική. Αυτά όλα είναι αντικείμενο συντονισμού. Εκεί υπάρχει συνδυασμός, εκεί υπάρχει κοινό τόπο, κοινή δομή, όπως είπε και ο Βάλτεμαρ. Οπότε πολλές φορές έχουμε χωριστές αποστολές με χωριστή εντολή για βάσιμους λόγους. Άρα χωριστή ιεραρχία αλλά κοινή δομή για, για τον συντονισμό και την υποστήριξη. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις ε, ξεκινώντας από την Αθηνά και την διαθεσιμότητα των κοινών κονδυλίων και αν μπορούν να βελτιώσουν την χρήση των δυνατοτήτων που έχουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι πολύ γρήγορα περνάμε στην ε, ταξιαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μονάδες αυτές, ε, τη γνωστή ιστορία, πολλές συζητήσεις από την στρατιωτική σκοπιά. Εμείς λέμε ότι είναι επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω από τη στρατιωτική σκοπιά είναι πλήρως λειτουργικό, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι έτοιμο για κρίση και αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το πρόβλημα είναι... Το πρόβλημα δεν είναι στο στρατιωτικό κομμάτι. Νομίζω ότι πιθανώς όταν μιλάμε για την κοινή χρηματοδότηση μπορεί να βελτιωθεί και ελπίζω επειδή οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται και η Επιτροπή της Αθηνάς εργάζεται σκληρά ε, επί των νέων προτάσεων ε, που μπορούν να διευρυθούν. Όπως ξέρετε, όταν μιλάμε για τους σχηματισμούς μάχης, ε, χρησιμοποιείται η κοινή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και όχι για όλες τις επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ευρύτερους τομείς που θα καλύπτονται π.χ. στρατηγία, επικοινωνίες, αυτές είναι κάποιες ιδέες και ελπίζω να βελτιωθεί έτσι η διαθεσιμότητα που νομίζω αυτό ήταν το ερώτημα του κυρίου Ζέμκα για του Ευρωπαϊκού στρατού ίσως να μην ήταν ξεκάθαρο έχουμε αυτές τις μονάδες ε, μάχης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό το κομμάτι ας πούμε αυτό που έχει αναπτυχθεί σε κάποιες χώρες ε, χρειάζεται η διοίκηση για να ενώσει όλες αυτές τις δυνατότητες και να τις χρησιμοποιήσει για ένα κοινό σκοπό. Ελπίζω λοιπόν να λειτουργήσει. Όταν μιλάμε τώρα για την εμπειρία και την διάκριση μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας. Πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει μια κοινή στήριξη και συντονισμός, αλλά συμφωνώ ότι αυτή η διάκριση μεταξύ βεβαίως πολιτικής και στρατιωτικής πτυχής τόπου είναι πολύ σημαντική, όπως βλέπουμε π.χ. όταν μιλάμε στις επαφές με τον ΟΗΕ. Θέλουν να μιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν να μιλήσουν με τον ΝΑΤΟ. Και εξετάζουμε διαφορετικές επιλογές. Οπότε πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση. Όταν μιλάμε για τις σχέσεις ε, μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Ε, ξεκάθαρο, κοιτάξτε, ο κεφαλής πολιτικής αποστολής είναι αρμόδιος για το πολιτικό σκέλος και τη στρατιωτική αποστολή για το στρατιωτικό. Βεβαίω ε, απαιτείται συντονισμό. Αυτό είναι το σκεπτικό. θέσα το ζήτημα των κοινών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, κάτι το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει βεβαίω να υπάρχει ε, συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο να χρησιμοποιηθούν ακριβώς αυτά τα οποία βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν μιλάμε τώρα για τις δυνατότητες ή την έλλειψη δυνατοτήτων που θέλουμε αναφέρθηκαν. Ακριβώς αυτή η στρατηγική πολλαπλασιαστές Παραδείγματος χάρη ένα αερίος ε, ανεφοδιασμός, ε, θαλάσσιες περιπολίες. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις απαιτήσει, ε, λίγο πολύ τα ίδια αναζητάμε με το ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση αυτή το θέμα της ΠΕΣΚΟ θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια λύση για το μέλλον. Για να βελτιωθούμε εδώ πέρα. Για τις ε, ΚΠΑ. Επίσης, όταν μιλάμε για τα στρατηγία, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πέντε κράτη-μέλη που προσφέρουν ε, επιχειρησιακά στρατηγία, ε, παρά το ότι έχουν όνομα επιχειρησιακά, είναι σε στρατηγικό επίπεδο. Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία. Έχουμε λοιπόν κάτι. Σχεδόν έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Ε, σχεδόν. Γιατί ε, σε καθημερινή βάση είναι άδειο. Είναι απλά υποδομές ε, έτοιμες να δεχτούν προσωπικό και να ενεργοποιηθεί το επιχειρησιακό στρατηγείο για μια αποστολή. Η λύση η οποία προτάθηκε με την εφαρμογή του NPCC είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία μόνιμη λύση. Δηλαδή όταν θέλουμε ακριβώ να ξεκινήσουμε την αποστολή η όλη διαδικασία ξεκινάει για πρώτη φορά ε, ζητάμε ποιο είναι, θα μπορούσε να είναι το προσωπικό και μετά ε, Βεβαίω η αναθεώρηση γιατί αναζητούμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μόνιμο και Βεβαίω, όταν μιλάμε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, μιλάμε για μια μόνιμη δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής για όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. για τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το τελευταίο θέμα να μην υπάρχει η αλληλεπικάλυψη. Κοιτάξτε, οι δυνατότητες ε, σχεδιασμού είναι 31 άτομα, ε, εκ των οποίων οι μισοί έχουν δύο ιδιότητες. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία ε, αλληλεπικαλύπτονται. Συγκρίνεται αυτό με το ΣΕΙΠ, το στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό παραδείγματο χάρη χρειάζεται 100 άτομα Όπω είχαμε στην Σομαλία 100 άτομα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Θα υπάρξει δεύτερο γύρο τραπέζη, ο κ. Μπούχνερ. His comments, myself as well. Ο κ. Μπούχνερ και εγώ θέλουμε να σχολιάσουμε. <clears throat> Okay. Ευχαριστώ. Όταν ε, αναφέρετε αυτές τις δομές, mm. τα ακουστικά, τα ακουστικά Ναι, όταν αναφέρετε αυτές τις δομές, έχω κάποια προβλήματα, γιατί σύμφωνα με τις ε, συνθήκες στην Ευρώπη και στην πράξη, τελικά, το Κοινοβούλιο δεν έχει καθόλου λόγο. σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας. Τώρα, όταν έχουμε λοιπόν νέες δομές με νέες ιεραρχίες, τότε το δημοκρατικό έλλειμμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Ε, έχουμε λοιπόν, κοιτάξτε, επί της αρχής ε, αποφάσεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να γίνονται από το Κοινοβούλιο, έτσι. Κάτι το οποίο εδώ πέρα δεν γίνεται. Um, uh, Το δικό μου σχόλιο, κύριε Νάβαρχε, είναι... Αν οι μικρές ή οι μεγάλες ε, δομές χρειάζονται και ένα νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν τα λειτουργικά θέματα, τα νομικά θέματα Υπάρχει και το θέμα του πώς ε, έχει αυτή τη δομή, της μορφής της δηλαδή, μορφή με μικρά γράμματα. Αυτή είναι και η ανησυχία μου, ότι πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και τις διπλές λειτουργίες εδώ και εκεί. Αλλά και νομικός πώς. Uh, also the we have to explore in... Αυτό πρέπει να το δούμε να το διερευνήσουμε ότι... και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι επικαλύψεις. Νομίζουμε ότι κλείνουν τώρα οι παρεμβάσεις. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Ακούω πάρα πολλούς τεχνικούς όρους, νομικούς όρους, ορολογία. Και στο μεταξύ αυτό που βλέπουμε στον πόλεμο στη Συρία, Φερρυπίν, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι η απόλυτη έλλειψη ευρωπαϊκής παρουσίας και δέσμευσης. Δεν υπάρχει κάτι που ήθελα και ζητούσα από τότε που έγινε Ευρωβουλευτής. Μια στεναρή σίγουρη για τον εαυτό της ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που να βασίζεται στη δύναμη που έχουν τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε αυτή την Ήπειρο, στην οικονομική δύναμη που έχουμε, που, που επηρεάζει πάρα πολύ για να χαλιναγωγήσει όλες αυτές τις δυνάμεις στη, στη Συρία ε, που κάνουν αυτόν τον πόλεμο δια αντιπροσώπου. με τρομερό ενδιαφέρον να σας ακούω, ε, γοητευμένος θα έλεγα, σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει, ε, τι να συντονίσουμε, ούτως ώστε να μην να παρισφρεί η μία, ο, ένας φορέας στα χωράφια του άλλου, ε, όλοι όσοι, όσοι φορείς ας πούμε δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, καλά όλα αυτά και άγια. Αλλά κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό από όλα είναι είναι ένας άνθρωπος που θα μιλήσει εκπροσωπώντας όλη αυτή τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απευθυνθεί σε αυτούς που αποφελούνται, που βγάζουν κέρδος από τον πόλεμο στη Συρία. Γιατί μέχρι το 2015 δεν είχαμε συνειδητοποιήσει καν ότι γινόταν πόλεμος εκεί πέρα. Μόλι, μέχρι να δούμε τις ε, πρώτες ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, προσφύγων στις πόρτες μας τότε συνειδητοποίησαμε ότι κάτι τρέχει στη γειτονιά μας. Φλιαρώ τώρα εγώ. Εσείς είσαστε οι εμπειρογνώμονες για να μου βρείτε λύσεις, προτάσεις και να τελειώσετε και τις φράσεις μου. Θα, θα θέλατε αγαπητοί κύριοι να σχολιάσετε. Βεβαίως θα καταγράψουμε τα σχόλιά σας. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε στρατιωτικός διοικητής. Σίγουρα δεν μπορώ λοιπόν να, σχολιάσω πολλά πράγματα. Μπορώ να τα διαμηνήσω στο Γενικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης απλώς. Σε σχέση με το αρχικό σημείο του κύριου Μπούχνερ. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για τις δομές. Ε, αυτό είναι το θέμα που μου δόθηκε. Ε, το θέμα της α, ανάπτυξης δεν αλλάζει το ποιος έχει την ευθύνη, τα κράτη-μέλη. Ε, και το MPCC είναι διαφορετική, εκεί υπάρχει διαφορετική αλυσίδα διοικητικό μηχανισμό, εν ε, η δομή είναι αυτή που αλλάζει. Η διοίκηση δεν αλλάζει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σχολιάσω τις πολιτικές ερωτήσεις. Εμείς οι στρατιωτικοί, όπως είπατε και εσείς, ασχολούμαστε με τα τεχνικά στοιχεία και εκεί θα παραμείνω στο τεχνικό, στην τεχνική σφαίρα. Εμείς δεν ε, ισχύζουμε ότι κάνουμε σχέδια προόπτου λειτουργικά 100% αλλά για τις ε, βασικές στρατιωτικές επιλογές που έχουμε και το πώς ε, τις εξετάζουμε ακριβώς για όλες τις περιοχές και θέατρα κρίσεων. Και η διοίκησή μας θα αξιολογήσει αυτά τα σχέδια, μπορεί να λειτουργήσουν, αξίζει να επενδύσουμε. Γιατί, και επιπλέον, θα χρειαστούν και επιπλέον έξοδα, γιατί εμείς κάναμε ένα αρχικό, μια αρχική εκτίμηση. Και όταν περάσουμε από το πλαίσιο της διαχείρισης των κρίσεων, περνάμε στην εφαρμογή, μετά πάμε στο κόνοψ, μετά πάμε στο σχέδιο πάρα πολύ προσπάθεια που γίνεται μετά από αυτή τη δική μας. Πριν όμως ληφθεί η πολιτική απόφαση, εμείς ετοιμάζουμε τα σχέδια. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το έργο μας και η αρμοδιότητά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Ναύαρχε, έχουμε απόλυτη συνείδηση των ορμοδιότητων σας, της αντολής σας. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας στη συζήτηση αυτή. Πολύ ενημερωτικά όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Και με αυτά νομίζω ότι κλείνουμε και αυτό το σημείο της ημέρησιας διάταξης. Θα ήθελα ακόμα μία φορά εκ μέρους όλων μας να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλό Πάσχα προφανώς. Ήταν το τελευταίο σημείο. Το τελευταίο ουσιαστικό σημείο. Έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Ερωτήσεις. Όχι. Και επομένως, να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 3 και 4 Μαΐου. Μια σημαντική πληροφορία. Έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να καλωσορίσουμε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Και να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία της μέσιας διάταξης. Καλό Πάσχα ακόμα μια φορά και θα ήθελα εδώ να κλείσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους πάντες, τη Ματία, τους Διερμηνείς. Καλό Πάσχα και από εμά. Γεια σας.